So, ladies and gentlemen, let's start. Um, Ας ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι που καθυστέρησα, πήγα σε λάθος αίθουσα. Σε άλλο κτίριο κιόλας. Συγγνώμη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως το πρώτο σημείο στην ημέρα διάταξη αφορά την ίδια τη σημερινή. Σχόλια, αλλαγές. Αν δεν έχετε κάποιο σχόλιο, πάμε κατευθείαν στο 2. Έγκριση των πρακτικών. Παρατηρήσεις, όχι. Πολύ ωραία, πάει και αυτό. Και μετά πάμε στο 3 ανακοινώσει Προέδρου. Ε, μιας και καθαρίσαμε Ας πάμε στο 4. 4. Εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Να δώσω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο Αγμό Ντεζόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω την έκθεση, την έχετε λάβει. Να σας πω που βρισκόμαστε με τις τροπολογίες να ευχαριστήσω τους διάφορους σκιώδεις που χρήσιμα συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της έκθεσης. Είχαμε καρποφόρες συνεδριάσεις και ευχαριστώ τον κύριο Πιτσουλά, Ραντός, Βαν Όρντεν, άλλος που συνέβαλαν καθοριστικά στον εμπλουτισμό της έκθεσης. Είχαμε τις τροπολογίες και προτείνω να τις ομοδοποιήσουμε σε 7 συμβαστικές για να ρυθμίσουμε κάποια ζητήματα. Μετά βεβαίως θα αποφασίσουν και θα αποφανθούν και οι ομάδες για τις επιμέρους τροπολογίες. Θα ήθελα να πω ότι οι τροπολογίες τηρούν τη φιλοσοφία της έκθεσής μας. Δηλαδή, μεταξύ δύο Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Δεκέμβρης 13 Ιούνις 15 για την ασφάλεια και την άμενα σε ένα πλαίσιο πολύ ανησυχητικό όσον αφορά την ασφάλεια και την άμενα επειδή όπως λέει και η έκθεσή μου νομίζω ότι 15 χρόνια το περιβάλλον μας δεν είχε τόσο έτσι ανησυχητική εικόνα όσον αφορά την ασφάλεια. Οπότε είναι υποχρέωσή μας να στείλουμε ένα μήνυμα λέγοντας ότι απέχουμε πολύ από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες μέλη συλλογικά σε επίπεδο Συμβουλίου. Βρισκόμαστε λοιπόν πολύ μακριά αλλά και ταυτόχρονα να είμαστε και επικοδομητικοί λέγοντας ότι θα πρέπει να εκλογικεύσουμε τις δεσμεύσεις μας. Βεβαίως υπάρχουν και διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με το βαθμό δέσμευσης που επιτρέπει η Ένωση. Αλλά τέλο πάντων κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί σήμερα ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί δεν βρίσκονται στο έξω των περιστάσεων και ότι ιδιαίτερα σε λειτουργικό επίπεδο αυτό που έχουμε στην Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αντικείμενο εκλογήκευση σε λειτουργικό, δημοσιονομικό, επιμελητιακό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προτεραιότητές μας και να παρεμβούμε ανάλογα. Χαίρομαι λοιπόν που η τεράστια πλειοψηφία των τροπολογιών ακολουθούν αυτή την φιλοσοφία, βεβαίως ξαναλέω με τις αποχρώσεις της κάθε, της της κάθε πολιτικής ομάδας. Αυτά από μένα, δεν έχω άλλα σχόλια να σας κάνω και ελπίζω να έχουμε την ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ το Μάρτιο νομίζω στο Στρασβούργο ώστε να έχουμε ένα τελικό κείμενο και ένα σημείο που αφορά τον τύπο. Εγώ δεν ήθελα να αποδεχτώ να υιαθετήσω σε αυτή τη φάση τροπολογίες που αφορούν την, τις πρώτες παραγράφους, τις αγωγικές δηλαδή, που αφορούν και παρουσιάζουν αυτή την φιλοσοφία. Δεν ήθελα λοιπόν να υιοθετήσω ή να αποδεχτώ τροπολογίες που είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς. Ξέρω ότι διάφοροι συνάδελφοι ήθελαν ενδεχομένω να αναπτύξουμε περισσότερο ας πούμε, τα θέματα όπως Ουκρανία, απειλή τρομοκρατίας. Αντίθετα θέλησα να μείνουμε έτσι πιο γενικόλογοι και να μην αναφερθούμε λεπτομερώς σε όλες τις κρίσεις γιατί μιλάμε για μια έκθεση που αφορά το σύνολο της πολιτικής άμυνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα πρώτα σχόλια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ κύριε Πίκουλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία. Κάνατε πολύ καλή δουλειά. Μας δώσατε ένα έγγραφο συνολικό, ένα έγγραφο διαρθρωμένο. Πολύ καλά σε ένα θέμα το οποίο έχει γεννήσει πολλά ερωτηματικά παρά έχει δώσει απαντήσεις. Έχουν κατεθεί τροπολογίες, συμβαστικές. Έχουμε καταθέσει και εμείς. Χαίρομαι που πολλές από τις ε, τροπολογίες της δικής μας ομάδας έχουν συμπεριληφθεί ε, στην έκθεση. Κάποιες ίσονος σημασίας μόνο παρατηρήσεις έχω. Πιστεύω όμως ότι θα συμβάλλουν στην ε, ποιότητα. Συμφωνώ με την γενική αξιολόγηση ότι πρόκειται για ε, καταγραφή της διεθνούς κρίσης και των κινδύνων για την ασφάλεια της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές λοιπόν και μακροχρόνιες ε, προκλήσεις και το περιβάλλον της Ένωσης δεν είναι ασφαλές. Η ασφάλεια μάλλον της δεν είναι σταθερή. Άρα λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο για την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια με όλα τα προβλεπόμενα δυνατά μέτρα. Θα θέλαμε μια πιο καλή και ισορροπημένη διατύπωση στις, ε, στην παραγράφο 11 για τις ε, αποστολές που θα έχουν πολιτικό, μη στρατιωτικό δηλαδή χαρακτήρα. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το φάσμα της διαχείρισης κρίσεων και των σχετικών παρεμβάσεων. Είναι καλά ισορροπημένη παραφός 18 τώρα όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών σε στρατιωτικές αποστολές και που είναι πιο σύμφωνη με την παράγραφο 21. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλέσει τα κράτη-μέλη να δείξουν περισσότερη βούληση για συνεργασία σε στρατιωτικές αποστολές και συμβολή στην ενίσχυση του δυναμικού που χρειάζεται. Το μόνο έκρεμες για μένα και αμφισβητούμενο ζήτημα, πώς ε, πρέπει να διαμορφωθεί η θέση της ΚΕΠΑ σε αυτήν την περίπτωση της κοινή ε, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, πώς θα διατυπωθεί και πώς θα συγκριθεί με τη σχέση μας με τον ΝΑΤΟ, παράγραφος 33 συγκεκριμένα. 22 είναι τα κοινά μέλη με την ε, συμμαχία αυτή, με την οργάνωση αυτή ασφαλείας και θα πρέπει να διατυπώσουμε πιστεύω όρους για την διαφάνεια όσον αφορά τη συμμετοχή και τη δράση τους. Κλείνοντα θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο, αλλά και όλους τους άλλους συνάδελφους που συνέβαλαν στην ε, έκθεση. Είναι πολύ καλά διαρθρωμένη, είναι εκτεταμένη και την υποστηρίζω πλήρως. Ευχαριστώ. Thank you. From um, Alde, I think it's Mr. Nard. Νάτ από την Alde. Ευχαριστώ. Εξ του κύριου Και εγώ να και κάποια δικά μου σχόλια. Ο κύριος Τράντος, σκιώδης, λέει ότι το κείμενο είναι ένα κείμενο συνενετικό και ισόρροπο. Θα ήθελα όμως εκτάκτως να πω ότι όσο δεν έχουμε μια καθορισμένη στρατογική ε, στρατηγική δράση που έχουν μόνο Γαλλία και Βρετανία, βρισκόμαστε στο πεδίο της ρητορική και της υποκρισίας. Και η αποστολή, οι ασκήσεις, οι στρατηγικές ασκήσεις στο Μάλι δεν ξέρω κατά πόσο επιτυχής είναι τη στιγμή που δεν έχει εγκατασταθεί καμιά στρατιωτική δύναμη εκεί. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε αμυντικές ασκήσεις, θα σας πούν όλοι οι στρατηγοί του κόσμου ότι είναι περιττό αυτό. Πάντως θα διατηρήσω τις εξαιρέσεις που ανέφερα, γιατί θεωρώ ότι αν δεν έχουν χώρες μέλη ένα σαφή στρατιωτικό ορισμό, θα εξαρτώμαστε πάντοτε από τους Άγγλους και τους Γάλλους, ενώ οι υπόλοιπε χώρε κάνουμε το πολιτικό σορθό, το οποίο είναι τίποτα. Thank you very much. Um, I have to... Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη. Μίλησε η ECR πριν από την Άλντε. Ελπίζω ο Τζέφρι να μην ανησυχήσει ακόμα περισσότερο. Ο Τζέφρι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω. Μια και η έκθεση δεν είναι τόσο κακή όσο περίμενα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συνειδητοποιούμε όλο και πιο πολύ ότι υπάρχει χρήσιμη ουσία σε αυτή την πολιτική. Ναι, πράγματι. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι του Άλντε, έχει κάποια χρησιμότητα η κρίση στην Κεντρική Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή υπογραμμίζουν την ανάγκη νότας δημοκρατίας και την εντόπιση κινδύνων από τους Ευρωπαίους και Ατλαντικούς συμμάχους πρέπει όλοι μας να λάβουμε υπόψη μας και να πάρουμε σοβαρά τις υποχρεώσεις μας για την άμυνα. Μιλήσαμε για την ανάγκη ταπάνης ε, τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ από τα μέλη του ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια ελάχιστη υποχρέωση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μην φανταστείτε ότι επειδή γίνονται εδώ συνεδριάσεις και υπάρχουν έγγραφα αυτό αρκεί. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο το ΝΑΤΟ έχει αξιοπιστία και αυτή η πολιτική νομίζω στην ουσία παρεκκλίνει από αυτό. Ανέκαθεν έλεγα ότι εδώ έχουμε ένα έτσι άκακο πολιτικό χόμπι σε δύσκολους σε εύκολους καιρούς. Τώρα όμως οι κύριοι έχουν γίνει δύσκολοι και προκλητικοί. Ελπίζω το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις και να εστιάσει τις προσπάθειες της Ένωσης σε πολιτικές δραστηριότητες που θα αφορούν βεβαίω τι δραστηριότητε του ΝΑΤΟ και τι χώρε μέλη και να ενθαρρύνουν τι χώρε μέλη να δράσουν όσον αφορά τα θέματα τη άμυνα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Κυρία Λέζινγκ δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Η Γκουέ έχει κάποιον που θέλει να λάβει το λόγο. Κυρία Σεμπάλος, πράσινη. Πρόεδρε, θα μιλήσω σου ειδικά για αυτό. Καλό να περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σα. Ξεκινάω ευχαριστώντα τον εισηγητή. για την πολύ καλή συνεργασία και τις χρήσιμες ε, συνεδριάσεις με τους κοινωνικούς που μπορούσαμε να καταλήξουμε σε χρήσιμες ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Θα συμφωνήσουμε με τους προγραλίσαντες Είμαστε ικανοποιημένοι από σχεδόν ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης. Ορισμένα μονοθέματα ε, δεν μας βρίσκουν 100% σύμφωνος. Θα πρέπει βεβαίως αυτό να το διευκρινίσω. Παράγραφη 6 και 25 επί παραδείγματι, εκεί που γίνεται λόγος για αυτονομία, στρατηγική αυτονομία. Νομίζω ότι είναι πολύ ασαφής όρος αυτός. Ε, θα έλεγα ότι είναι ακόμη και επαναστατικός μέχρι πυρηνικού δυναμικού. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι η ανάπτυξη των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας Όταν λέμε αυτονομία όμως, είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αυτές οι αξίες. Ευχαριστώ πάντως τον εισηγητή που δέχθηκε την παραπομπή στο άρθρο 21 της Συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Δεν έχουμε καταλήξει στο θέμα αυτό της στρατηγικής αυτονομίας πώς θα ψηφίσουμε. Για την παράγραφο 11. Η διατύπωση των πολιτικών εργαλείων, των μη στρατιωτικών αποστολές αποστολών συγγνώμη, ε, δεν είναι πολύ σαφή, ιδιαίτερα με την έμφαση που δίνεται κατά την παράθεση στις στρατιωτικέ αποστολέ. Εν πάση περιπτώσει, για μας, η στάση μας θα κριθεί και από την πρόταση που αφορά εθνικά κοινοβούλια, εθνικούς προϋπολογισμούς. Το 2% δεν νομίζω ότι καλύπτει ξεκάθαρα την ιδέα της ποιότητας της άμυνας που προσφέρεται. Περισσότερο έχει ποσοτική χρειά. Και τώρα λέμε να ορίζουμε το 2% είναι σαν να ενθαρρύνουμε τις αρχές στα κράτη-μέλη να αρχίσουν να τα, να διασκορπίζουν τα χρήματα των φορολογουμένων σε τέτοιου είδους δαπάνες. Δεν υπάρχει λόγος να αγοράζουν εξοπλισμούς. Ξέρουμε ότι υπάρχει υλικό σε μεγάλη ποσότητα. Αεροσκάφη, τεθωρακισμένα που δεν αξιοποιούνται. Και αυτά αποτελούν απλώς εσπάθηση των χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογημένου ή των εθνικών φορολογημένων. Θέλουμε λοιπόν ποιοτική αναφορά και όχι ποσοτική. Θέλουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να συμπηλήσουν ποιοτικό υλικό αξιοποιώντας καλά τα χρήματα του φορολογουμένου. Με όρους όμως ποιοτικούς και όχι ποσοτικούς. Και πιστεύουμε ότι επιπλέον μέσα και πόροι που ενδεχομένως ε, περισσεύουν θα πρέπει να πάνε στην πρόληψη. 200 δις ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο για την άμυνα. Φτάνουν αυτά. Όχι μόνο φτάνουν, αλλά θα μπορούσαν και να περιοριστούν οι σχετικές δαπάνες με συνεργασία των ε, ένοπλων δυνάμεων και γενικά ε, του κλάδου της άμυνας μεταξύ των κρατών. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε και στο άρθρο 31. Δεν θέλουμε σχέδια για ανάπτυξη ε, μη επανδρομένων, ευρωπαϊκών μη επανδρομένων αεροπλάνων. Γι' αυτό υποστηρίζουμε το 123, εκεί που λέμε ότι χρειάζεται η ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για τα μη επανδρομένα αεροπλάνα. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μη επανδρομένων που θα σημαίνει ουσιαστικά ότι τα κράτη-μέλη μεμονωμένα θα συμβάλλουν, θα συνεισφέρουν στην ε, εκτός ε, ενόμου τάξεως εκτέλεση αποφάσεων όπως συμβαίνει σε σχέση με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, παραδείγματι, πλευρά των ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ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 Θέλω να ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την έκθεση. Έρχεται εν ευθέτω χρόνο μεταξύ των δύο ε, συνόδων κορυφής για την άμυνα και νομίζω ότι εμείς ως Ευρωβουλευτές καλούμεθα να αξιολογήσουμε την κατάσταση τέσσερις μήνες λίγο πριν από την προσεχή σύνοδο κορυφής να δούμε σε σχέση με τα όσα αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο του 2013 τι έχει συγκεκριμένα εφαρμοστεί τι προχωρεί προς εφαρμογή και τι ακόμη δεν έχει καλυφθεί. Άρα θα πρέπει να επισημάνουμε τα σημεία στα οποία παραμένουν κάποια ελλείμματα ακόμα, εκεί που θα πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση. πίεση. Θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι πριν από μερικές εβδομάδες συνέβησαν γεγονότα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν στην ορθή τους διάσταση, υποβιβάστηκαν, υποβιβάστηκε η σημασία τους. Ε, αυτό δεν μας βοηθάει. Θέλω να φερθώ και σε ένα σημείο που ακούστηκε από συναδέλφους, αυτό που αφορά τη στρατηγική αυτονομία. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία δεν στρέφεται εναντίον κανενός συγκεκριμένα. Έχει σημασία όμως αυτή η, η στρατηγική αυτονομία. Διότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι πάντοτε θα μπορούμε αυτομάτως να αντλούμε την υποστήριξη των δυνάμεων και των πόρων του ΝΑΤΟ. Γιατί μπορεί οι Αμερικανοί να μην θέλουν να συμπράξουν. Ή γιατί κράτη μη ε, που δεν ανέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά ανήκουν στο ΝΑΤΟ, έξι τον αριθμό, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία σημειώνω, μπορεί να μην θέλουν να συμπράξουν. Επί παραδείγματι, η Τουρκία μπορεί να μην θέλει για λόγου πολιτική περιφερειακή σε σχέση με τόσα συμβαίνουν στο Ιράκ ή σε άλλο κομμάτι του ε, μουσουλμανικού κόσμου να μην θέλει να συμπράξει. Μπορεί να έχει άλλε επιλογέ. Δεν αποκλείεται αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν εμεί να εξαρτώμεθα ω Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από την αξιοποίηση των πόρων του ΝΑΤΟ και από ένα πιθανό βέτο. Αυτή η στρατηγική λοιπόν αυτονομία νομίζω αποτελεί ένα μέτρο προληπτικό ούτω ή ε, δεδομένων των φιλοδοξιών μας ως Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην χρειάζεται να εξαρτώμεθα από το ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο έχουμε ε, περιγράψει ως ελλείμματα ως ελλείψεις στην πολιτική μας και καταγράφονται στην έκθεση. Νομίζω ότι δεν αρκεί να το καταγράφουμε, πρέπει να προχωρήσουμε σε προτάσεις για λύσεις. Επί παραδείγματος το security of supply, ασφάλεια προμηθειών. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να το καταγράψουμε όπως έγινε με το Δεκέμβριο του 2013 και να λέμε ότι να υπάρχει ένα φαινόμενο και θα το διαπιστώνουμε σε κάθε αντίστοιχη κατάσταση. Όχι. Υπάρχει μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε θέση να διαπιστώνουμε αν μπορεί ο βιομηχανικός κλάδος, ε, ο αμυντικός κλάδος να καλύπτει τις ανάγκες και αναλόγως, εάν δεν τις καλύπτει, να συμπληρώνουμε τα κενά. Σε αυτό θα ήθελα εγώ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και όπω υπόθηκε και στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή των Προϋπολογισμών, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση, τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού Αθηνά. Γιατί αυτή τη στιγμή όπω έχει πραγματικά εμποδίζει την αποτελεσματική δραστηριοποίησή μα, Είτε γιατί είναι overcharged ή overstretched, δηλαδή είναι στο όριο των δυνατοτήτων του ή έχει ξεπεράσει το όριο των δυνατοτήτων του, ή γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα 100% χρηματοδότησης των ε, δράσεων. Παράδειγμα, η Ελλάδα έχει η εχει ξεπερασει τα πολλά καράβια, δυνατοτητα 100 χρηματοδοτηση των πάρα πολλά αεροπλάνα αλλά χρήμα δεν έχει. Άμα λοιπόν μιλούμε για την ανάπτυξη μιας ναυτικής επιχείρησης, με τον εφιστάμενο μηχανισμό θα έπρεπε να υπάρξει μια ομόφωνη απόφαση ποιος θα το πράξει αυτό, διότι ξέρετε ότι ασφαλώς οι Έλληνες φίλοι δεν θα μπορέσουν να συμπράξουν, θα πούνε πλοία έχουμε αλλά δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την επιχείρηση. Άρα λοιπόν με τη μεταρρύθμιση ενός μηχανισμού Αθηνά που θα φρόντιζε και για την καταγραφή ποσο, μιας κλίδας ποσοστιαίας κατανομής ανάλογα με τα κράτη. Θα αξιοποιούσαμε αυτά που υπάρχουν στη θέση μας. Θα ρωτούσαμε την κυρία Μογκερίνη, θέλουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Θα ρωτούσαμε τους Έλληνες, θα μας λέγανε έχουμε καράβια. Θα ρωτούσαμε τους Πορτογάλους, θα μας λέγανε έχουμε καράβια. Και μετά, ανάλογα με, το, με τη συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, το 2-3% θα συνέβαλαν και το υπόλοιπο θα το πλήρωναν οι υπόλοιποι. Ιδιαίτερα διαφορετικά θα έπρεπε να βγουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, όποιο άλλο έχει πλοία και 100% να δεσμευτεί σε μια τέτοια επιχείρηση. 100%. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και πρέπει να το εξηγήσουμε στους ε, ομολόγους μας βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Να τους εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ο πιο σωστό δρόμο. Και βέβαια να, να επισέλθει και η οικονομική αυτή διάσταση. Ευχαριστώ κύριο Σαφοζέχ.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 ότι αυτή η συμμαχία είναι συμμαχία πολέμου. Δεν είναι αλήθεια. Νομίζω το δεύτερο ήμιση του περασμένου αιώνα δεν είχαμε κάποιο πόλεμο στην Ευρώπη, οπότε δεν συμφωνώ. Το έγγραφο αυτό, η έκθεση, πρέπει να παρουσιάζει τις γενικές μας θέσεις για αυτή την πολιτική. Όμως, όμως για να έχει κάποιο νόημα, πρέπει να παρουσιάσουμε και εμείς τις επιμέρους θέσεις μας για την πολιτική αυτή. Γι' αυτό σας ενθαρρύνω στις τροπολογίες σας να περιλάβετε μία παραπομπή, μία μνήα σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας. Μιλάω ας πούμε για τροπολογίες που αφορούν πυρηνική ενέργεια, επίδειξη δύναμης από την Ρωσία μελή της Ένωσης που και αυτό δεν έχουν. Καταλήξη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε μια κοινή προοπτική ασφάλειας, θα πρέπει αυτή η προοπτική να είναι εκτρώνουν κάνε φόρος. Εάν θέλουμε να επιτύχει, θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να βρουν τη θέση τους μέσα στην έκθεση αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη πρέπει να σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, να μεριμνούμε για το πιο αδύνατο, για το πιο ευάλωτο. Και επίσης, όταν μιλούμε για συνεργασία, στον αμυντικό κλάδο. Η Ευρώπη απέχει πόρο από μια οικονομική συνοχή. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πορεία και η εικόνα των λιγότερο ευμερουσών οικονομιών και των αμυντικών τους κλάδων. Θα ήθελα ένα έγγραφο το οποίο θα μιλάει σε δύο διαστάσεις, δηλαδή πρώτα στη διάσταση της ε, αλληλεγγύης και δεύτερον στην ε, πράξη, στα πραγματικά ζητήματα, στα αληθινά ζητήματα, ώστε να μην ε, αναφερόμαστε σε αφηρημένες ελπίδες ότι κάπου πολύ μακριά βρίσκεται και μια Ευρώπη. Ευχαριστώ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 et euh, ainsi euh, les euh, actions que nous devons mener à l'extérieur de l'Union στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών. Στο πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να επιμείνουμε για την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών μας υπηρεσιών πληροφοριών ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε προληπτική δράση καλύτερη από ό,τι μέχρι σήμερα. όχι μόνο στο ευρωπαϊκό έδαφος, όπως το είδαμε αυτό ήδη στην Γαλλία και στη Δανία πρόσφατα, αλλά και προς το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε προληπτική δράση, όπου υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες. Ε, υπάρχει λοιπόν η πρόταση του Μάτιο Ρέντσι για τη δημιουργία μας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών. Είναι παράξενο σήμερα μόνο τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτούν μια υπηρεσία ε, πληροφοριών που είναι στα πρώτα της βήματα από τη στιγμή που θα έχουμε διάσκεψη κορυφής για την άμυνα που θα οργανωθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, πρέπει να πραγματοποιήσουμε κάποιες μελέτες για να συνοδεύσουμε αυτές τις προτάσεις ε, στο επίπεδο το ευρωπαϊκό που έγιναν από τον Ματέο Ρέντσι. Ακόμη, έχουμε, πρέπει να έχουμε μία σχέση με το Μισελ Μπαρνιέ που διορίστηκε από την Κομισιόν επικεφαλής μιας αποστολής για την ασφάλεια και την άμυνα. Και σε αυτό το τομέα των πληροφοριών ε, ήρθα σε επαφή μαζί του πρόσφατα και μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή την επαφή ώστε να οδηγηθούμε ε, σε μια ενισχυμένη άμυνα και ασφάλεια στην Ευρώπη λόγω των απειλών. Πρόεδρος. Τελειώσαμε λοιπόν τα σχόλια. Ο εισηγητής. Ε, κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας, το οποίο αντανακλά αυτό το οποίο έλεγα στην αρχή, δηλαδή επικοδομητικό πνεύμα από όλους, βάσιμα σχόλια στη μεγάλη τους πλειοψηφία, σχόλια τα οποία σέβομαι απόλυτα όσον αφορά την πολιτική τους νομιμοποίηση ο Μίκελ Γκαλόρ. Ε, μου αφαίρεσε από το στόμα, αν θέλετε, ορισμένα επιχειρήματα για ένα θέμα το οποίο έχει γίνει κλασικό θέμα στις συζητήσεις μας. Ο Τζέφρι Τζόρνταν δεν είναι εδώ, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για την άρθρωση με τον ΝΑΤΟ, Εβραίος. Το ΝΑΤΟ λοιπόν δεν μπορεί, δεν θέλει και δεν πρέπει να κάνει τα πάντα. Θα έλεγα ρεαλιστικά λοιπόν πέραν από οποιαδήποτε ιδεολογία μπορούμε να διαπιστώσουμε το εξής. Σε όλα τα πεδία κρίσης που εμφανίζονται το ΝΑΤΟ δεν πρέπει, δεν θέλει και δεν κάνει, να κάνει τα πάντα. Η Ευρώπη πρέπει λοιπόν να παίξει το ρόλο της. Τώρα πρέπει να προσδιορίσουμε το ρόλο της. Μια Ευρώπη με λίγα κράτη-μέλη, μια Ευρώπη που κάνει συμμαχία αυτών που θέλουν ή τι. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση. Το ότι επαφιόμεθα απόλυτα στο ΝΑΤΟ στρατιωτικά δεν έχει νόημα, διότι υπάρχουν χώροι κρίσης που το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να πάει, δεν θα θέλει να πάει και οι επιτόπου δεν θα θέλουν επίσης να πάει. Προσπαθήστε να το κάνετε αυτό στην Αφρική, στο Μαλή. Καλή δύναμη, δεν θα γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, ε, δεν πρέπει κάτι να γίνει για το κέρας της Αφρικής, για το Μαλή. Λοιπόν, έξι χώρες μη ευρωπαϊκές είναι μέλη του ΝΑΤΟ υπάρχει πολύ ισχυρή, αλλά και οι υπόλοιπε πέντε που έχουν προβληματικούς πολιτικούς προσανατολισμούς. Ο Μικαέλ αναφέρθηκε ήδη στην Τουρκία. Αν σήμερα θέλετε να οργανώσετε μια επιχείρηση στην Βόρεια Αφρική με στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεν θα μπορέσετε διότι θα πέσει βέτο από την Τουρκία. Αυτές είναι αλήθειες που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας για να αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε μια αυτόνομη ικανότητα της Ευρώπης που δεν είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ αλλά θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Ε, το άρθρο 42 της των συνθηκών είναι σαφέστατο. Τώρα, όσον αφορά την στρατηγική αυτονομία, τυπικά είναι πάντα θέμα συζήτησης. Αυτή η έκφραση ε, πάντοτε περιλαμβανόταν ε, στις εκθέσεις μας. Και μπορούμε βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι ε, αυτονόητο επιχείρημα ή εξατομικευμένο, αλλά σημαίνει την ικανότητα της Ευρώπης να πει ναι ή όχι για κάποιες επιχειρήσεις τις οποίες δεν θα έθελε ή ήθελε να αναλυφθούν εκ μέρους της. Θετικά ή αρνητικά αυτή η αυτονομία ε, έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Ας πάρουμε το Ιράκ. η αρνητικα αυτη η αυτονομια εχει τη δυνατοτητα να εκφραστει ας παρουμε το ιρακ ρακινή περιπέτεια των Αμερικανών ε, το 2003 είναι ακριβώς το να πει κανείς όχι σε μια τέτοια περιπέτεια. Η αυτονομία σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε σε μέρη που άλλοι δεν μπορούν να πάνε και εκφράζεται και πολιτικά και στρατιωτικά. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή τη φιλοδοξία. Είναι περισσότερο μια φιλοδοξία παρά μια αλήθεια, αλλά πρέπει να την υποστηρίξουμε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το 2%. Μπορεί να μοιάζει περίεργο για ορισμένους, αλλά συμφωνώ μάλλον με το επιχείρημά σας. Ο απόλυτος στόχος του 2% στο ΝΑΤΟ είναι ποσοτικός στόχος που δεν λαμβάνει υπόψη του τις ποιοτικές προσπάθειες ορισμένων χωρών. Η θέση της Γαλλίας πάντα ήταν όχι ταμπού για το 2%. Ας εξετάσουμε καλύτερα τι γίνεται όσον αφορά τις επενδύσεις και την έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι πιο σημαίνοντα από ένα 2% του ΑΕΠ που είναι απόλυτα ποσοτικό μέγεθος και που άλλωστε μπορεί να οδηγήσει σε λάθος ερμηνείας όσον αφορά τις πραγματικές αμυντικές προσπάθειες των κρατών. Αν δείτε ποιος φτάνει στο 2% σήμερα, θα δείτε ότι δεν είναι αυτοί που συμβάλλουν περισσότερο στη βιομηχανία της άμυνας και στη στρατηγική. Η τροπολογία Van Merden είναι αυτή η οποία προσφέρει περισσότερη ευληγησία για αυτό το θέμα, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται. Και θα ήθελα να την υποστηρίξω. Όσον αφορά τα μη επανδρομένα. Βεβαίω, όλοι ονειρευόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για τη χρησιμοποίηση των μη επανδρομένων πτήσεων. Ε, δεν ε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια νομοθεσία δικιά της που δεν θα είναι επιχειρησιακή και δεν θα περιληφθεί σε ένα ευρύτερο νομικό πλαίσιο παραδείγματο χάρη στον ΟΗΕ. Και υπάρχει περιθώριο χρονικό προς το παρόν, διότι Όσον αφορά τα προγράμματα των μη επανδρομένων πτήσεων, ε, έχουν προοπτική 20 ετών και προτού φτάσουμε στη δημιουργία των μη επανδρομένων πτήσεων που μπορούν να στοχεύουν όπως τα αμερικανικά ή οι αμερικανικές, ε, έχουμε χρόνο. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, Βεβαίως ε, θα δεχθούμε την τροπολογία του ειδικού επί του θέματος στην υποεπιτροπή μας. Ε, δεν επεκτάθηκα πάνω στο θέμα γιατί ήξερα ότι θα παρέμβεις. Ε, υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων και σου αφήνω την πατρότητα αυτής της τροπολογίας που είναι πλήρης και σημαντική. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μικέλ Γκαλέρ όσον αφορά την χρηματοδότηση τη ΕΠΑ που κατά την άποψή μου ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση αλλά δύσκολα θα υποστηριχθεί από το Συμβούλιο. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα του μηχανισμού Αθηνά και γενικά των ικανοτήτων. Ε, μου κάνει εντύπωση που μέσα στο ΝΑΤΟ οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να αποκτήσουν εξοπλισμό από κοινού χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ και οι ίδιες χώρες που θα θέλανε μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο από κοινού να αποκτήσουν εξοπλισμό δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτό δεν κολλάει με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ανάπτυξη των ικανοτήτων μας. Ε, ε, ε Σόφχαουζερ. Έχουμε διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει ε, να καταδικάσουμε την πολιτική άμυνα στην κοινή βάση της επικουρικότητας. Ε, μιλάμε για διακυβερνητική πολιτική. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι τα κράτη-μέλη τα οποία αποφασίζουν σε αυτό το τομέα και τελικά η δυνατότητα των κρατών μελών είναι αυτή η οποία προσδιορίζει τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό. Το θέμα λοιπόν της επικουρικότητας εξορισμού περιλαμβάνεται στην υπόθεση που εξετάζουμε. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ επανέρχομαι. Πάντα με ανησυχεί ε, η αντιαμερικανική στάση του πολιτικού σας ε, σχηματισμού. Δικιά σας η ευθύνη βέβαια, μπορούμε να το συζητάμε ώρες. Αλλά εγώ δεν είμαι άτομο που λέω ναι ναι ναι στις πολιτικές θέσεις της Αμερικής. Αλλά και το τελείως αντίθετο οδηγεί στο παράλογο και αυτό με ανησυχεί στις συζητήσεις μας. Όσον αφορά τα πυρηνικά Βεβαίως και υπάρχουν πυρηνικές απειλές στα σύνορά μας, έτσι τις αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απαφίεται είτε στο ΝΑΤΟ ή στο δόγμα των κρατών μελών που είναι πυρηνικές δυνάμεις. Και γι' αυτό δεν αναφερόμαστε στην έκθεση σε αυτό το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποια μέρα να ανοίξουμε τη συζήτηση πάνω στο πυρηνικό ζήτημα. Αλλά όπως έχουν σήμερα τα δόγματα, τα αμυντικά, δεν εμπίπτει η αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφοριών, ήταν το τελευταίο σχόλιο και θα καταλήξω με αυτό. Αμφιβάλλω και ε, είμαι προσεκτικός. Ε, ε, η διατύπωση του Ρέντσι για μία CIA ευρωπαϊκή, τι να πω, ε, οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι αποτελεσματικές, λειτουργούν σωστά, έχουν νομοθετικό πλαίσιο, επιχειρησιακό πλαίσιο, συγκεκριμένο, συγκεκριμένο στην κάθε χώρα. Η συνεργασία δεν απαγορεύεται, είναι διακριτική, εμπιστευτική, απόρριτη, αλλά αυτό δεν σοκάρει περσέ, αυτή είναι η φύση του πράγματος και η θέληση να αποκτήσουμε ε, μια, έναν υπερφορέα ευρωπαϊκό δεν θα φέρει κατά την άποψή μου αποτελεσματικότητα. Οι υπηρεσίες ζητούν συνεργασία. Δεν ζητούν ένα υπερφορέα ευρωπαϊκό. Ε, έχω μεγάλες επιφυλάξεις πάνω σε αυτό. Έχω πάντα την τάση να μην καταλαβαίνω την ε, υπεραξία αν θέλετε ενός τέτοιου φορέα. Έχουμε μια intelligence agency στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ε, συμμερίζονται όλες τις πληροφορίες όσον αφορά την τρομοκρατία. Ο φορέας αυτός προσφέρει μια πλατφόρμα ανταλλαγών πολύ ενδιαφέρουσα, ε, έχει καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών, διατίθενται ενδιαφέρουσες πληροφορίες εκεί και δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ διότι ε, προτού δημιουργήσουμε αμοιβαία συμμετοχή στην πληροφορία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε την πληροφορία. Και οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι αυτές που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βεβαίως η ρευστότητα, η ροή μάλλον των πληροφοριών μπορεί να βελτιωθεί. Ε, νομίζω ότι έχω αναφερθεί λίγο πολύ σε όλα τα θέματα που θέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Um, äh, Ευχαριστώ, Αγνώ. Πριν το κλείσουμε και νομίζω ότι θα είναι σημαντική συμβολή της υποεπιτροπής μας για τη συνεχιζόμενη συζήτηση. Θυμάμαι πάντα ε, μια φράση ενός διπλωμάτη από την ε, Σύνοδο ασφαλεία του Μονάχου που έλεγε ότι μπορεί οι Γάλλοι να είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν αλλά όχι να πληρώσουν, οι Γερμανοί να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αλλά όχι να πολεμήσουν και οι Βρετανοί να μην είναι διατεθειμένοι να κάνουν οτιδήποτε από τα δύο. Αυτό ε, σε ένα πιο ελαφρύ τόνο και ζητώ συγγνώμη. 9 Μαρτίου λοιπόν πάει στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων, Ολομέλεια 1η του Απριλίου. Κλείνουμε έτσι το θέμα για να περάσουμε αμέσως στο επόμενο που αφορά την ενημέρωση σχετικά με την αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η U4RCA ολοκληρώνει την ε, αποστολή της εκεί. Είχαμε τον Αγνόντο Ντοζό, είχαμε τον κύριο Παγνού, κύριο, την κυρία Καμπάλος, εκτός από την κυρία Φωτίγκα. Θέλουμε λοιπόν... Ε, μια και δεν είναι εδώ η Πρόεδρος. Να μας ε, εξηγήσει ο Αγνό Ντονζάν. Ναι, μια και έχω προθερμάνει τη φωνή μου, συνεχίσω. Ε, βέβαια θα μιλήσει και ο κύριος Βαγνιό και η κυρία Σεμπαλός. Μέλη και εκείνη της αντιπροσωπείας μας υπό την κυρία Φωτίγκα, την Πρόεδρο. Αυτές τις ε, τελευταίες χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είχα την ευκαιρία πρέπει να πω να επισκεφθώ σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις και αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ήταν μια αποστολή πολύ καλά ε, οργανωμένη, επιτυχέστατη, την οργάνωσε και η δική μας η γραμματεία και η επιτόπου αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία και ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή. Στη χώρα αυτή δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για με τον όρο χώρα. Εν πάση περιπτώσει το κράτος αυτό που βρίσκεται σε μια δυσχερέστατη κατάσταση, μάλλον για failed state πρέπει να μιλούμε, δηλαδή αποτυχημένο ε, κράτος και αυτό ήταν και ο πρώτος στόχος της ε, αποστολής, να διαπιστώσουμε την κατάσταση και τη συμβολή της U4RCA. Ε, πρέπει να πω λοιπόν ότι ήμασταν αρχικά πολύ επικριτικοί εναντί αυτής της επιχείρησης όμως ομολογώ ότι ολοκλήρωσε τον στόχο, το στόχο της που ήταν από τον Απρίλιο του 2014 στον Πάγκη να διασφαλίσει κάποια σημεία στρατηγικά το αεροδρόμιο πρώτα που τώρα έχει μεταφερθεί στον έλεγχο των Εθνών και δύο ε, περιοχές περιφέρειες του Μπάγκη, παριθμών 3 και 5 που είχαν τα περισσότερα προβλήματα ασφάλειας. Η αποστολή με 750 περίπου άτομα από 10 διαφορετικές χώρες και συμμετοχή σημαντική τρίτων κρατών, ε, Γεωργίας και Σερβίας συγκεκριμένα, λειτουργήσε αποτελεσματικά. Συναντηθήκαμε με τη διοίκηση και το προσωπικό της αποστολής και όλοι έδειξαν κάτι το συνηθισμένο και κάτι που γίνεται και συστηματικά σε τέτοιες αποστολές, την ε, συστηματική αυτή δουλειά, την αναλυτική αυτή δουλειά, την καλή αυτή δουλειά που κάνουν ε, άντρε και γυναίκε που συμμετέχουν σε αυτέ τι αποστολέ και θα ήθελα να του ευχαριστήσω. Η αλυσίδα τη διοίκηση φαίνεται να λειτουργεί κατά τρόπο ικανοποιητικό και πρέπει να σημειώσω ότι αυτό δεν είναι πάντοτε δεδομένο σε αποστολέ οι οποίε έχουν κατά, την, ε, κατά το σχεδιασμό των συμμετεχουσών δυνάμεων τέτοιου είδους προβλήματα. Πάντως εδώ φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά. Η διάρθρωση με άλλες παρούσες δυνάμεις, τις δύο συγκεκριμένα, ε, της Αγκαρής από τη Γαλλία, που ήταν η πρώτη που αναπτύχθηκε, και τις δυνάμεις Μινούσκα των Ηνωμένων Εθνών, με 10.000 περίπου άντρε. και τη μεγαλύτερη κατά πάσα πιθανότητα ετερογένεια, αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό των δυνάμεων του ΟΗΕ. Ήτανε καλή. Η U4 κλείνει, τα μαζεύει το Μάρτιο, 15 Μαρτίου και Εδώ τίθενται ερωτήματα ως προς τη μετάβαση, δηλαδή πώς θα γίνει η μεταφορά στις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών του έργου που προηγουμένως επιτελούσε η UFOR και ποια θα είναι η αποδοχή από τις τοπικές αρχές, ε, τους πολίτες αλλά και τους λοιπούς διεθνείς φορείς θα μπορέσει δηλαδή με την ετερογένεια που χαρακτηρίζει και που μερικές φορές αποτελεί και μειονέκτημα ε, του ΟΗΕ ε, να υποκαταστήσει στο έργο της τη UFOR. Πρώτο ερώτημα. Άλλα ερωτήματα είναι αυτό της παρουσίας και τη στράτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να έχει παρουσία με πολύ πιο περιορισμένες δυνάμεις και εντολή περισσότερο παροχή συμβουλών η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην αναμόρφωση των ενόπλων δυνάμεων της Κεντρικής ε, Αφρικής, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια αποστολή όμως η οποία δεν έχει μπορέσει να ολοκληρωθεί. Οι οδύνες είναι πολύ ε, μακροχρόνιες για την παραγωγή της. Ε, το προσωπικό που έχει ζητηθεί μόνο κατά το 1 τρίτο προσφέρεται και δι' από τη Γαλλία μόνο. Ε, από αυτά που βλέπουμε υπάρχει δυσκολία λοιπόν, δυστοκία, αλλά και δυσκολία ως προς την αντίληψη της αποστολής και της σημασίας της. Δηλαδή έχουν την εντύπωση και οι αρχές και οι πολίτες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ότι θα πάει αυτή η αποστολή πιο περιορισμένης ε, εμβέλειας να κάνει την ίδια αποστολή που είχε και τη U4 ή αντίστοιχες ε, δράσεις με αυτές που είχαν οι δυνάμεις μας στο Μαλί και ε, στη Σομαλία όπου ε, είχαν αναλάβει την εκπαίδευση των ανώπλων δυνάμεων. Πρέπει λοιπόν αυτό καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν είναι ε, επαρκές το προσωπικό. Παραμένει προς το παρόν αυτή η αποστολή όπως σας είπα με τα ερωτηματικά της. Πρέπει να δούμε αν είναι καταρχάς καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνει τέτοιο έργο. Μου λένε βέβαια αν δεν το αναλάμβανε η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο, ε, πραγματικό το ερώτημα και σοβαρό διότι δεν είμαι... Αλλά από την άλλη δεν είμαι και πεπισμένο ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύονται εν ώψη αυτής της κρίσης, οι αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε, ναι, αλλά συμφέροντα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που αποτυγχάνει στη λειτουργία του ένα κράτος που γίνεται failed state, δηλαδή θα αναλαμβάνει δράση. Και μια δεύτερη ερώτηση που σας δεν τολμώ να θέσω, αλλά ε, δίνω απάντηση χωρίς να την έχω θέσει. Η παρέμβαση ήταν ε, κατά βάση γαλλική ως προς τη σύνθεση, ως προς την έμπνευση. Επιτυχής βέβαια. Και επί τη ευκαιρία συγχαίρω τους ε, Γάλλους στρατιωτικούς που έλαβαν μέρος στην αποστολή αυτή. Είναι όμως δυνατόν να συνεχίζουμε να στέλνουμε ευρωπαϊκές αποστολές που βασικά είναι γαλλικές με χρώματα ευρωπαϊκά. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να μας απασχολήσει και άλλωστε αυτό συνδέεται και με το προηγούμενό μας ζήτημα, τα δημοσιονομικά δηλαδή προβλήματα, γιατί υπήρξαν χώρες που μας ε, ε, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή, χώρες όμως να έχουν τα απαραίτητα μέσα. Άλλες χώρες οι οποίες έστειλαν προσωπικό ε, αξίζουν συγχαρητηρίων, έστω και με τις περιορισμένες δυνατότητες που είχαν. Για τους Ισπανούς Φερρυπίν που θέλω ρητά να αναφέρω, το μηχανολογικό επίσης της Ιταλία είχε πολύ σημαντική προσφορά, όσο περιορισμένη ε, αξία τεράστιας. Και για να κλείσω υπογραμμίζω ότι ναι είχα επικριτική στάση στην αρχή αλλά διαπιστώνω πολύ σημαντική ε, ε, είχα πολύ επικριτική στάση όμως διαπιστώνω ότι η U4RCA είχε πολύ σημαντική επιτυχία κλείνοντας. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Ναι παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Η παρουσίαση που έγινε ήταν ενδιαφέρουσα. Αλλά εμένα το θέμα αυτό με έχει απασχολήσει πολύ. Και αυτοί που έχουν εργαστεί στην EUFOR είχαν εκφράσει ανησυχίες για το τι θα γίνει μετά την αγχώρηση της ΕΟΦΟΡ και την ανάληψη των καθηκόντων αυτών από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη λοιπόν είπαν ότι έχουν την ικανότητα, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα καθήκοντα της ΕΟΦΟΡ. Οπότε προς το παρόν δεν ανησυχώ. Νομίζω ότι η δουλειά που ξεκίνησε θα μπορούσε κάλλιστα να συνεχιστεί και βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Νομίζω ότι όταν θα βρεθεί η κατάλληλη στιγμή για την άναξη της επιχείρησης, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη στιγμή για το κλείσιμο της επιχείρησης. Όμως, δυστυχώς, η κατάσταση ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η επιχείρηση αυτή, λοιπόν, εξελίσσεται. Αν θέλουμε, λοιπόν, να πετύχουμε τους στόχους μας, θα πρέπει εμείς ε, να εμπλακούμε και μέσω της κοινωνίας των πολιτών για την επικοδόμηση της χώρας αυτής, ανοικοδόμηση της χώρας αυτής και την ανάπτυξή της. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο το να πάμε σε αυτή τη χώρα, να κάνουμε αυτή την επιχείρηση και μετά να φύγουμε και να τα αφήσουμε όλα όπως ήταν πριν. Δεν τα βοηθήσουμε και πολύ έτσι. Θα πρέπει να δώσουμε ένα νόημα και μια αξία στις πράξεις μας, αλλιώς θα είναι περιττές. Επίσης έχουμε και το θέμα των διακρίσεων όσον αφορά τις δυνάμεις που παρεμβαίνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να το συζητήσουμε ώστε να υπάρξει και μια συμφιλίωση των διαφόρων ομάδων που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και που είναι σημαντικό να γίνει. Και αυτό δεν αφορά μόνο την θρησκεία αλλά και την φιλετική καταγωγή. Αυτά είναι δεσμεύσεις για το μέλλον που δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό σκέλος γιατί αυτή η πεπατημένη δεν είναι η μοναδική. Ευχαριστώ. Ναι, συνάδελφοι, πρόεδρε, πολύ σύντομα. Μετά από τον απολογισμό τον λεπτομερή και κέριο του συναδέλφου Ανώ και μετά από αυτό που είπε η κυρία Σεμπάλιος, να πω μόνο τα εξής, συμπληρωματικά κι εγώ. Να έχουμε κατά νου ότι αυτή η κατάσταση όπως τη γνωρίζουμε σε αυτή τη χώρα σχετίζεται με ένα πολιτικό πλαίσιο που σχετίζεται και αυτό με τη σειρά του με την τρομοκρατία σε αυτή την περιοχή. Κοντά στο Μπαγκί υπάρχουν γιατί υπάρχουν μόνο 600 χιλιόμετρα απόσταση μεταξύ του θέατρου των επιχειρήσεων και του Μπαγκί, δηλαδή όπου εμπλέκεται το Τσάντ, το Καμερούν και η Νιγηρία, κατά του Μπόκο Χάραμ. Ο διοικητής της γαλλικής δύναμης μας έλεγε ότι λίγες μέρες πριν την αφεξή μας υπήρξαν χριστιανοί οι οποίοι είχαν πάει στα βορειοδυτικά στα σύνορα με το Καμερούν οι οποίοι απήχθησαν και δολοφονήθηκαν από τη Μπόκο Χάραμ μια ομάδα που συνδέεται με την Μπόκο Χάραμ. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και το λέω αυτό προς τον συνάδελφο. Μήπως η Ένωση λοιπόν θα έπρεπε στα πλαίσια αυτής της επιχείρησης να λάβει υπόψη της και τέτοια συμβάντα. Εγώ νομίζω ναι, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ζητήματα καθαρά εσωτερικά της Κέντρο Αφρικανικής Δημοκρατίας, αλλά έχουμε να κάνουμε θέματα γενικότερα ασφάλειας που αφορούν ολόκληρη την περιοχή ή την υποπεριοχή τέλο πάντων. Εδώ ακριβώς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τρομοκρατίας που πλήττουν ε, συμφέροντα ευρωπαϊκά και όχι μόνο γαλλικά. Εδώ λοιπόν μια πρώτη απάντηση δίνω για τη χρησιμότητα αυτής της αποστολής. Δεύτερο σημείο, το είπε και ο Αρνό και ο Μποντήλ, του EU4 στις 17 του Μάρτη θα αποχωρήσει, θα μπορούσε να αντικατασταθεί, όχι ακριβώς να αντικατασταθεί, αλλά τέλος πάντων ε, θα έχουμε ε, στρατηγικούς συμβούλους Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε γιατί ο στρατός δεν υπάρχει πια της κεντροαφρικανικής ε, δημοκρατίας. Υπάρχουν 6.000 άντρες οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά εκεί σε κάποια στρατόπεδα αλλά οποίοι όμως είναι άοπλοι κοντά στον πάγκι. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς εμείς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην αναδιάρθρωση αυτού του στρατεύματος χωρίς να πούμε ότι εντάξει εμείς δουλέψαμε για ένα χρόνο, τελειώσαμε, φύγαμε και δεν μας νοιάζει τι γίνεται μετά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι το μέλλον αυτής της χώρας εξαρτάται με την συνολική μας πολιτική για τα εξωτερικά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπως είπε και ο συνάδελφος είναι και θέμα χρηματοδότησης. Εμείς, η Ευρώπη, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ε, αναδιάρθρωση του στρατού της χώρας αυτής αλλά και της οικονομίας. Αλλά θα πρέπει να συμμετάσχουν και η διεθνή κοινότητα, ο ΙΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του κλπ. Τρίτον, Υπάρχει επίσης και η ανάγκη η Ένωση να συνεχίσει να αναπτύσσει πολιτικές ανθρωπιστικής βοήθειας, όχι μόνο μέσω της Επιτροπής μας για την άμυνα, και να αναπτυχθεί μια πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχέση με αυτούς τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολίες όπως έλεγε η Μποντήλ. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε την παρέμβασή μας. Και τέλος, τελευταίο σημείο, να πω ότι πολιτικά η ανοικοδόμηση αυτής της χώρας με εκλογές σε πρώτη φάση, μετά σύνταξη συντάγματος, με εκλογή προέδρου στη συνέχεια που προς το παρόν προβλέπονται για τον Αύγουστο, αλλά ίσως να είναι ανεπαρκής αυτός ο χρόνος, οπότε ίσως να πάμε το φθινόπωρο το 16. Η Ευρώπη λοιπόν δεν θα πρέπει να μείνει ξένη όσον αφορά την διοργάνωση προεκλογικών εκλογών σε αυτή τη χώρα γιατί θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα από τους κύριους πυλώνες της ανικοδόμησης της χώρας και της ασφάλειας όμως στο σύνολο της υποπεριοχής ενώπιον και σε σχέση με την Μπόκο Χάραμ όπως έλεγα προηγουμένως 43 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για τις ευρωεκλογέ. Συμφωνώ με τον Αρνό λοιπόν που έλεγε ότι Κάθε φορά γίνεται το ίδιο. Η Γαλλία χρηματοδοτεί. Σήμερα έχουμε λοιπόν 19 εκατομμύρια που βρέθηκαν μόνο σε εισαγωγικά. Αλλά ως ποσό είναι ανεπαρκές για την διοργάνωση αυτών των προεδρικών εκλογών που αποτελεί ένα πέρασμα υποχρεωτικό, μια μετάβαση υποχρεωτική προς την σταθερότητα της χώρας αυτής. Θα σας υπενθυμίσω, αγαπητές συνάδελφοι, ότι είναι παρόντες οι εκπρόσωποι που θα μας κάνουν την παρουσίαση, γι' αυτό θα σας παρακαλώ να είναι σύντομη η παρέμβασή σας, κύριε Νάρτ. Δεν υπάρχει κεντροαφρικανική δημοκρατία. Η αποστολή στον Μπάγκη αφορούσε το να αποτρέψουμε να συνεχίσει να αποτελεί ένα κέντρο ολέθρου το μπάγκι για τους μεν και τους δε. Μιλώντας λοιπόν για την ανοικοδόμηση του στρατού, πρέπει να λέμε πρώτα ότι πρέπει να ε, ανοικοδομήσουμε ένα συμβασμό μεταξύ των φυλών για να δούμε μετά ποιος θα απαρτίζει το στρατό. Από την Ταρούγκα μέχρι το Μπάγκι, τα ανατολικά δηλαδή της χώρας, η περιοχή αυτή βρίσκεται εκτός ελέγχου το δυτικό τμήμα τελείως διαφορετικό. Αλλά έχουμε προβλήματα με τον έλεγχο αυτών των περιοχών. Οπότε όταν συζητήσουμε για εκλογικές διαδικασίε, για προεδρικές εκλογές, για μια πολιτική υπερδομή τη στιγμή που η εθνική και η κοινωνική δομή στη χώρα αυτή δεν υπάρχει καν, αυτό σημαίνει ότι είμαστε αυτάρισκοι και ότι δημιουργούμε μια κενή δομή η οποία δεν ανταποκρίνεται σε απολύτως τίποτα. Ο πρόεδρος Μποσισέ υποστηρίχθηκε από το Τσάτ και μετά τον κατέστρεψαν μέσω μιας διαδικασίας που αφορά ολόκληρη την ανατολική, ανατολική περιοχή της χώρας που είχαν πια αποφασίσει να απορρίψουν την κυριαρχία των φυλών, των τόπιων φυλών. Οπότε εμεί δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη ρητορική τη χώρα, αλλά θα πρέπει να, βρούμε, να συμβάλλουμε στο να βρεθεί μια συνένεση. Οπότε πριν από το στρατό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη συνένεση που δημιουργεί το ίδιο το κράτο και μετά ο στρατό. Οπότε υπό την άποψη αυτή οι προεκλογικέ συγγνώμη, οι προεδρικέ εκλογέ δεν αποτελεί τίποτα παρά ασκήσει επιχάρτου που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Και έτσι κλείνει το σημείο αυτό τη σημερινή διάταξη. Εξ ονόματος της υποεπιτροπής ορίζω τον αντιστράτεγο Γκί Μπουφσενσμιτ, διοικητή του Eurocor. Χρόνια τώρα η επιτροπή μας, η υποεπιτροπή μας συνεργάζεται στενά με το Eurocor. Ξεκινάω λοιπόν με μια πολύ σύντομη διατύπωση ερωτήσεων σε μια κατάσταση λίγο σταθερή, με προβλήματα στην ασφάλεια δηλαδή. Περιμένουμε, κύριε, α, μάλλον, στρατηγέ, Βόξον Σμιτ, να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα αναπτύσσει μια σημαντική αποστολή από την αρχή του καλοκαιριού, το Eurocore. Αναλαμβάνει εκπαιδευτική δραστηριότητα κατάρτισε στο Μαλή. Και αυτό είναι σημαντικό βήμα, το ότι ξεκινάει την εκπαίδευση των απλών δυνάμεων εκεί. Σημαντικό βήμα για την Eurocore, σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές είναι οι προσδοκίες από την αποστολή αυτή. Πάντα Πρόκληση μεγάλη βέβαια είναι για το στρατιωτικό, για τις ενόπλες δυνάμεις να εκφράζονται μεγάλες προσδοκίες από πλευρά των πολιτικών. Και με αυτή τη σύντομη σταγωγή σας δίνω το λόγο. Oh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Υποεπιτροπής, καλημέρα σας. Είμαι ο αντιστράτηγος Γκί Μπούσον Σμιτ. Είμαι Βέλγος και όχι Γερμανός. Η σύγχυση είναι συχνή λόγω του ονόματός μου. Έχουμε τα ίδια χρώματα με τη γερμανική σημαία αλλά ανάποδα και συχνά στο Στρασβούργο μου λένε μιλάτε πολύ καλά γαλλικά για ένα Γερμανό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε σήμερα. Δεν είναι κάθε μέρα που ο διοικητής της Eurocore μπορεί να μιλήσει σε ένα τόσο σημαντικό ακροατήριο. Δεν έχω επίσημη εντολή να σας μιλήσω. Συνεπώς, ό,τι θα σας πω σήμερα δεν καλύπτεται ούτε από την κοινή ηγεσία της Eurocore, ούτε από την ανώτατη ηγεσία του Βελγίου. Σας μιλώ σαν υπεύθυνο της Eurocore. Ε, ε, ε, έχω μια επιχειρησιακή εμπειρία και συγκεκριμένα εμπειρία στην κεντροϊκή Αφρική. Είμαι στρατιωτικός και όχι πολιτικός. Δεν θα τοποθετηθώ σε πολιτικά θέματα, όμως είναι ε, ιδιαίτερη δομή το Eurocore και συνεπώς έστω και αν εμείς οι στρατιωτικοί σκεφτόμαστε τα στρατιωτικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας επηρεάζει ο πολιτικός κόσμος, προσπαθούμε να καταλάβουμε τα όσα συμβαίνουν και να επηρεάσουμε και τις αποφάσεις βεβαίω. Λοιπόν, ήθελα να αρχίσω με μία παρουσίαση για το Eurocorp per se και στη συνέχεια να σας δώσω κάποιες ε, προσωπικές τοποθετήσεις για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Θα το αντιστρέψω. Θα ξεκινήσω να σας μιλήσω που έχουν για θέματα που έχουν περισσότερο να κάνουν με την ηγεσία, το γιατί και πώς και μετά θα σας παρουσιάσω τα slides, τις διαφάνειες για να σας δείξω πώς διοικείται το Eurocom. Ξεκινώ λοιπόν με κάποιες ιδέες, κάποιες προσωπικές σκέψεις ως προς την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Είμαι λίγο εικονοκλάστης, αλλά δεν περιμένετε να σας πω μόνο καλά νέα, φαντάζομαι. Πρώτο θέμα που θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, το στρατιωτικό δυναμικό στην Ευρώπη υπάρχει και είναι σημαντικό, αλλά παρακμάζει. Αναφερθήκατε στο 2% του ΑΕΠ, σε πολλά ε, κράτη δεν φτάνουμε εκεί και οπωσδήποτε το Βέλγιο δεν είναι το καλό παράδειγμα. Αυτό το οποίο με ανησυχεί σε αυτή την απεικοδόμηση του στρατιωτικού μηχανισμού στην Ευρώπη είναι ότι φτάνει μια υπογραφή ε, για να ε, διαλύσει κανείς ένα μηχανισμό, αλλά μπορεί από την άλλη πλευρά να χρειάζεται 10-20 χρόνια για να δημιουργήσει ένα μηχανισμό. Λοιπόν, απεικοδομούμε συνεχώς τις χώρες μας τον στρατιωτικό μηχανισμό. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι η διαδικασία λήψης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαρύς, ε, δίσκαμπτη. Θυμηθείτε το 2003 την επιχείρηση Άρτεμις στο βορρά του Κονγκό, στην περιοχή Αμπούνια. Εκεί οργανώσαμε μία επιχειρήση με κάποιες συμβάλλουσες χώρες, κυρίως η κυρίως η Γαλλία για τα στρατεύματα ξηράς και το Βέλιο για τις μεταφορές. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτή την επιχείρηση αποφεύγοντας κάποιους μηχανισμούς απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέτυχε η επιχείρηση. Αυτό καταδεικνύει ότι μπορούμε να πάμε επί τόπου και να ενεργήσουμε. Η συνένεση βεβαίω η ευρωπαϊκή σταματάει τη λήψη αποφάσεων. Και θα σας μιλήσω αργότερα για τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών. Όταν έχουμε λοιπόν 28 κράτη-μέλη, είναι <coughs> σχετικά δύσκολο να φτάσουμε σε συνέντευξη. Δίκο το Eurocore με έξι χώρες πλαίσιο όπου να είναι. Η συνένεση η καθημερινή δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι στα ημικύκλιά σας το να υπάρξει συμφωνία μεταξύ 28 χωρών για μία δράση είναι μία πρόκληση αξεπέραστη. Το θέμα λοιπόν της πολιτικής θέλησης με ανησυχεί. Δεν επικρίνω, διαπιστώνω. Είναι σαφές ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κάποια δυναμία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Αυτή η αδυναμία, αυτή η έλλειψη πολιτικής στέλσης, είναι προσωπική η ανάλυση που κάνω, εξαρτάται και από την κουλτούρα της Ευρώπης που βασικά ασχολείται με τη διπλωματία, τα δημοσιονομικά, την οικονομία. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα ενός βιβλίου του Μπερ Βεντρίν. Μπορεί να το μας αρέσει ή όχι, αλλά είναι ενδιαφέρον το απόσπασμα. Λέει, οι ευρωπαϊκοί λαοί θέλουν να πιστέψουν μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλου, Πόλεμο ότι η βία δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί. Καλό είναι αυτό, αλλά κάνουν λάθος. Αυτή η αντίληψη του κόσμου από τους ευρωπαϊκούς λαούς σε σχέση με την τοποθέτηση του ρεαλισμού, δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε τις ΜΚΟ και τους πνευματικούς ανθρώπους που θέλουν το καλό πράγμα και από την άλλη πλευρά έχουμε τους κακούς, δυτικούς εναντίον των υπολείπων. Είναι, εκφράζει παιδικότητα η οποία ουσιαστικά μας παραλύει διπλωματικά και πραγματικά. Πρόκειται για μια ηρεαλιστική πολιτική που είναι φλίαρη ε, δεν πλησιάζει τον ρεαλισμό καθόλου, είναι αδύναμη και δίνει ελπίδες για πράγματα ανέφικτα. Λοιπόν, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Οφείλεται αυτό σε διάφορους παράγοντες, δεν θα επεκταθώ. Δεν υπάρχει συνένεση όσον αφορά τα ζωτικά συμφέροντα και τις απειλές. Η Πολωνία ε, δεν μπορεί να βλέπει με τον ίδιο τρόπο την κέντρο αφρικανική δημοκρατία όπως ε, ε, η Γαλλία. Δεν μπορεί πούμε η Ουκρανία να γίνεται αντιληπτή από τις βαλτικές χώρες με τον ίδιο τρόπο όπως από άλλες χώρες. Συνεπώς είναι δύσκολο να έχουμε συνένεση, ομοφωνία για τα ζωτικά συμφέροντα αναφερθήκαμε στις δυσκολίες στο Μαλί. Το επίπεδο της ε, επιχείρησης ήταν σχετικά χαμηλό, εκπαίδευση των στρατιωτικών για αμυντική δράση αρχικά. Δεν πρέπει κανείς να είναι υπερφιλόδοξος εξ αρχής. Η εμπειρία μου μου λέει όσον αφορά την ανοικοδόμηση του στρατού στο Κονγκό ότι πρέπει κανείς να ξεκινάει από την αρχή. Μόνο όταν έχετε τοπικές δυνάμεις που είναι σε θέση να έχουν αμυντική δράση, μπορείτε να τις οδηγήσετε και σε επιθετική δράση που είναι πιο περίπλοκο. Είναι θέμα χρόνου. Δεν φταίνε οι στρατιωτικοί μας. Και σύμφωνο με τον κύριο Ντονζόν που αναφέρθηκε στις δυνάμεις της Γαλλίας στο Σαγκάρις, φαντάζομαι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, της υποστήριξης ε, της λογιστικής. Και όσον αφορά τον ε, Ευρωπαίο, νομίζω ότι ο Ευρωπαίος δεν έχει εκπαιδευτεί. Συνεπώς, έχει μία λάθος αντίληψη ασφάλειας μέσα στα σύνορα του Σέγγεν από καιρούς καιρών υπάρχει κάποιο συμβάν. Κοπενχάγη, Παρίσι κτλ. Αλλά μετά από δύο-τρεις εβδομάδες κάθεται πάλι σκόνη και ο Ευρωπαίος ξαναγίνεται καταναλωτής. Δεν υπάρχει κουλτούρα του Ευρωπαίου όσον αφορά την άμυνα, διότι δεν έχει σωστή αντίληψη των απειλών. Κι όμως αυτές οι απειλές υπάρχουν και φοβάμαι ότι η αφύπνιση θα γίνει τη στιγμή που εμείς οι Ευρωπαίοι στο σύνολό μας και κατά τρόπο συνεχή θα αντιληφθούμε την απειλή κατά των ζωτικών μας συμφερόντων. Είτε θα έχουμε ένα κράσ στα χρηματιστήρια, είτε τρομοκρατικές ενέργειες στα σύνορα, συνεχώς στα σύνορα του Σέγγεν, είτε θα απειλούνται τα συμφέροντά μας στο εξωτερικό, είτε θα απειλούνται τα πληροφοριακά μας δίκτυα στον κυβερνοχώρο, είτε θα έχουμε συμβατικές ε, στρατιωτικές απειλές. Πάρτε την Ανατολική Ευρώπη. Αφελώς πιστεύαμε ότι δεν θα χρειαζόταν να έχουμε ξανά σενάριο ε, συγκρούσεων. Βλέπετε όμως ότι δεν το γλιτώσαμε. Υπάρχει και κάτι άλλο που μας αποσταθεροποιεί, η ροή των λαθρομεναστών. Ε, έχουν περάσει πολύ καιρός και τώρα Έχουμε μετανάστες που φτάνουν κατά χιλιάδες και τίποτα δεν σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό θα σταματήσει καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται ε, εντατικά στην Αφρική. Αναφερθήκαμε εκτενώς προηγουμένως στο ρόλο του ΝΑΤΟ. Έχω μία μέτρια τοποθέτηση εδώ, διότι το, ε, το Eurocore είναι μια δομή που χρησιμοποιείται και από τον ΝΑΤΟ και από τον ΟΗΕ. Συνεπώς, γενικά συμφωνώ ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πανάκια και θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να εκχωρήσουμε την ασφάλειά μας στο ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανοί σαφέστατα δεν θα συνεχίσουν επαόριστο να υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Άμυνα και να αναλαμβάνουν τη δικιά μας την ασφάλεια. Θα επαναπροσωνατολίσουν τα συμφέροντά τους προς την Ασία, πιθανότατα μεταξύ άλλων. Συνεπώς, αυτή η βοήθεια η Αμερικανική και του ΝΑΤΟ, βασικά το ΝΑΤΟ είναι οι Αμερικανοί, αυτή η βοήθεια θα μειωθεί κάποια στιγμή και οι Αμερικανοί θα μας κοιτάξουν στα μάτια και θα μας πούν να αναλάβουμε τη δικιά μας την ασφάλεια μόνοι μας. Συνεπώς, συμφωνώ με όσους από εσά είπαν ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κάποια στρατηγική αυτονομία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ ασχολείται με τα στρατιωτικά και η ΕΕ ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα. Είναι λάθος αυτό. Ε, κάθε αποστολή βεβαίως εμπεριέχει μια στρατιωτική πτυχή και μια πολιτική πτυχή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε αποστολή στο εξωτερικό πρέπει να βασίζεται στα, στα τρία στηρίγματά της, την άμυνα, την ανάπτυξη και τη διπλωματία. Δεν είναι μια σαφώς στρατιωτική επιχείρηση και δεν είναι μια σαφώς διπλωματική επιχείρηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Σας θα δώσω ένα παράδειγμα, το Κονγκό. Ειδικότερα ήμουν υπεύθυνο για την αναδιάρθρωση των στρατευμάτων του Κονγκό. Η αναδιάρθρωση ήταν καλό πράγμα, αλλά έπρεπε να συνοδευτεί από συγκεκριμένες δράσεις στο διπλωματικό επίπεδο και στο αναπτυξιακό. Δεν είμαι κάποιος που θέλω πολέμους, προτιμώ όπως όλοι οι στρατιωτικοί να μην έχουμε πόλεμο, αλλά δεν πρέπει ε, να πιστεύουμε ότι υπάρχει απαλή δύναμη χωρίς ισχυρή δύναμη. Έστω και αν η Ευρώπη έχει χαμηλό προφίλ και βασίζεται στο ΝΑΤΟ και ε, βασίζεται στην έννοια της έξυπνης δύναμης, πιστεύω ότι θα βρεθούμε σε δυσκολίες μελλοντικά. Αυτά λοιπόν ήταν Αυτές ήταν ε, προσωπικές σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Άμυνη. Μην θεωρήσετε ότι είναι απεσιόδοξα όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν ε, ε, καλές ιδέες που πρέπει να υιοθετήσουμε και άλλες που πρέπει να απορρίψουμε. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι αυτής της παρουσίασης. Θα είμαι σύντομο. Το εργαλείο του οποίου έχω την τιμή να ηγούμε 28, από τις 28 Ιουνίου του 2013 και θα αφήσω τον Ιούνιο του 2015. Ξεκινώ λοιπόν δείχνοντα σα σε ποιο βαθμό το Eurocore είναι ένα εργαλείο συγκρίσιμο με τα άλλα επιτελεία ενόπλων δυνάμεων και πόσο μπορεί να είναι εναλλακτικό και συγκεκριμένο εργαλείο και σε ποιο σημείο έχει φτάσει στην πρόοδο και την ε, ύπαρξή του στο χάρτη αυτών που δεν έχουν οι διάθεσή τους έχετε το τις αρχές που υπάγονται στο ΝΑΤΟ με τα οικόσημά τους ξεκινώντας λοιπόν από Ράκη προς Ανατολάς βλέπετε την Βρετανική Βλέπετε το Στετίν της Πολωνίας, βλέπετε τη Γερμανική, βλέπετε τις μονάδες της Ελλάδας και της Τουρκίας, νοτιοανατολικά την Ισπανία, στο κέντρο Eurocore, γαλλικό σώμα και το γερμανό Ολλανδικό. Εννέα λοιπόν γενικά επιτελεία. Τι είναι το γενικό επιτελείο. Πρέπει να αποφύγουμε μία σύγχυση ο όρος Γενικό Επιτελείο Στρατού παραμένει ως όρος από τον ψυχρό πόλεμο. Ήταν δηλαδή ε, μία μονάδα η οποία είχε στη διάθεσή της 60.000 στρατιώτες και μπορούσε να προχωρήσει επιχειρήσεις. Αυτό δεν το κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για 60.000 στρατιώτες. Καμία δύναμη ευρωπαϊκή μόνη της, ακόμη και πολλές μεταξύ τους θα μπορούσαν να συλλέξουν στρατό 60.000 ανδρών. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε συνήθως στρατηγούς με τρία αστέρια επικεφαλής μιας μονάδας η οποία μπορεί να αναλάβει δράση σε ένα περίπλοκο σχετικά περιβάλλον. Αυτό λίγο πολύ είναι η έννοια των δυνάμεών μας. Αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πάρα πολύ και δείχνει το χωριό Eurocore σε μια επιχείρηση πριν από μερικά χρόνια. Δείχνει και το... την παρακαταθήκη, την ε, κληρονομιά ότως το field camping όπως το λέγαμε, αυτά που παραμένουν στη διάθεσή μας, στη διάθεση του Eurocore προκειμένου να αναπτύξουμε αυτή την πραγματική πόλη του Eurocore. Εδώ υπενθυμίζω ότι το Eurocore είναι μια δομή που αρχικά ήταν στη διάθεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Πριν από 23 χρόνια ιδρύθηκε ως εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκάτοχοί μου όμως πολύ γρήγορα αντελήφθησαν ότι θα πρέπει να αντιτεθεί και στη διάθεση του ΝΑΤΟ. Πολύ γρήγορα υπογράψαμε λοιπόν συμφωνίες με το ΣΑΚΕΡ, την Ευρωπαϊκή πτυχή του ΝΑΤΟ και επίσης αντελήφθησαν ότι πρέπει οι επιχειρήσεις που θα αναλαμβάνει το Eurocor να καθοδηγούνται από, τις, ε, είναι από τα Ηνωμένα Έθνη, υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ένα από τα πιο έμπειρα σώματα ενόπλων δυνάμεων. Από την ίδρυσή του πριν από 22-23 χρόνια έχει αναλάβει μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό το 1998 στη Βοσνία ριζεγοβινη το 2000 στην ε, πρώην Ιουκοσλαβία πάλι, στο Ίσαφ στη Αφγανιστάν, 300 ε, ε, σε δύο εναλλαγές το 2012 πάλι στο Αφγανιστάν, με διάφορες πτυχές, με διάφορες δομές και δύο φορές το ΝΑΤΟ μας χαρακτήρισε NATO Response Force ε, σήμα κατά τη του ΝΑΤΟ πολύ πολύ ζηλευτό. Για να σας δείξω καταρχάς το πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό το σώμα. Πριν από 22 χρόνια, όταν πρώτο δημιουργήθηκε, υπήρξε πρώτα η ταξιαρχία, η γαλλογερμανική. Ο πρώτος λοιπόν Μιτεράν και ο καγκελάριος Κολ είχαν την ιδέα για τη συγκρότηση του σώματος με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της απαραίτητης ευρωπαϊκής άμυνας. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του Eurocorps είναι η χρησιμότητά του. Ε, πρέπει να υπάρχει ένας διοικητής, ε, λέμε συνήθως αλλά δυστυχώς εδώ αυτό δεν ισχύει. Εγώ έχω ως ανώτερο αυτό που λέμε κοινή επιτροπή, δηλαδή ένα μη μόνιμο όργανο, το οποίο ακριβώς είναι υπεύθυνο ο επικεφαλής άμυνας και περιλαμβάνει τους ε, επικεφαλής των επιτελείων και τους ε, υπουργού αμήνης από χώρες πλαίσιο. Πέντε χώρες τώρα, έξι σε λίγο. Έχω λοιπόν δέκα ε, προϊσταμένους και ο διάδοχός μου θα έχει δώδεκα κάτι το οποίο δεν δυσκολεί τα πράγματα, αλλά πάντων. Τρίτο σημείο που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε το Eurocore ως ένα μοναδικό, ένα ενιαίο γενικό επιτελείο είναι αυτό που αφορά τη συνθήκη του Στρασβούργου που δίνει στο Eurocorps μεγάλη αυτονομία και οικονομική και δικαστική. Ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, εγώ θα πάω φυλακή. Έτσι. Να το έχει υπόψη με αυτό επόμενος θα το ανατρέξω γρήγορα αυτό, αλλά τόσο πάνω να σας δείξω ότι στην ε, πυραμίδα της ε, διαφάνειας θα δείτε ότι έχουμε την Κοινή Επιτροπή και έχουμε εδώ πέρα τέλο πάντων ένα, έτσι, ένα στερισμό διαφορών άλλων οργάνων και υπευθύνων αλλά τέλο πάντων δεν έχουμε ευρωπαϊκά πράγματα αλλά προσπαθούμε το περιβάλλον γνωστό, Στρασβούργο καταρχάς, το ξέρετε όλοι νομίζω δεν είμαστε μακριά από τα ευρωπαϊκά όργανα και επίσης έχουμε επαφή με πανεπιστημιακά όργανα πρώτης τάξεως, η ΕΝΑ και το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών, κάτι που οποίο μας επιτρέπει να έχουμε ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων και να διοργανώνουμε μαζί τους ε, ενδιαφέρουσες έτσι, εκδηλώσεις. Επόμενη διαφάνεια. Διάδροση Eurocore. Θα μου πείτε πού είναι ο στρατό σας. Δεν έχω στρατό. Κανείς διοικητή ε, σώματο στρατού δεν έχει στρατό. Έχουμε ένα γενικό επιτελείο με περίπου χίλιου άντρες και γυναίκες, πολίτε και στρατιωτικούς. Και έχουμε και μια βοηθητική ταξιαρχία, ταξιαρχία υποστήριξη. Τώρα, οι δυνάμει οι οποίε διατίθενται στο EuroCorp αυτέ ε, αναπερίπτωση παρέχονται. Αυτό ισχύει τώρα και αυτό αφορά την διαδικασία που στην ουσία αποτελεί μια πτέρνα όσον αφορά την λήψη των αποφάσεων, την εκτέλεσή του κτλ. Όσο η δομή ιεραρχία υπάρχει, ε, είναι εκπαιδευμένη και επιβεβαιωμένη, εντάξει, αλλά αν δεν υπάρχει, αν δεν ισχύει αυτό, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ιεραρχία διοίκηση. Οι χώρε, οι αρχικέ Γαλλία, Γερμανία ε, συνοδεύτηκαν μετά από Λουξεμβούργο, Ισπανία, Βέλγιο. Η Πολωνία θα προσθεθεί από το 2016 1η Γενάρη, έκτη χώρα πλαίσιο. Υπάρχουν εδώ Πολωνοί. Α, να, εδώ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε συμπατριώτες μας Πολωνούς στη δομή μας, επειδή νομίζω ότι συμβάλλουν με μια εναλλακτική πολιτική νοοτροπία, θαυμάσια συνήθω ποιότητα και ευχαριστώ πολύ την Πολωνία. Έχουμε λοιπόν τρει συνδεδεμένε χώρε οι οποίες ε, έχουν μειωμένα δικαιώματα, υπερισμένα δικαιώματα ε, τρεις Ιταλούς, δύο Ελλήνε, δύο Τούρκου. Η συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων λειτουργεί θαυμάσια εδώ σε εμά. Επόμενη, κάποια στοιχεία για τη συμμετοχή. Βλέπετε ότι η κάθε χώρα συμβάλλει με τα δικά τη μέσα. Αν δούμε το Βέλγιο, παρέχει 151 άτομα προσωπικό. Πολύ σημαντική συμβολή θα έλεγα κάτω δεξιά θα δείτε την Αμερικανική σημαία έστω και αν έχει ευρωπαϊκή υπόσταση αυτή η δομή δεν ξέρω τι θα ήταν καλό να έχουμε στην παρέλαση και Αμερικανική σημαία αλλά έχουμε βέβαια στην παρουσία της Αμερικής και στις δομές του ΝΑΤΟ αλλά και στη δομή εκπαίδευσης του σώματός μας. Οργανωτική δομή. Αυτή τη στιγμή ε, είμαστε έξι στρατηγοί στο Eurocorp. Έχουμε Βέλγος, έχουμε και Ισπανούς, ο αρχαίος επιτελείου είναι Γάλλος και μετά έχουμε άλλους τρεις ε, στρατηγούς ε, με ένα αστέρι για τις ταξιαρχίες, Βέλγο, Πολωνό, Γερμανό. Αυτό σας δείχνει ακριβώς την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα πλαίσια του Eurocorp, δηλαδή το μοναδικό γενικό επιτελείο σώματος στρατού, το οποίο είναι πραγματικά πολυεθνικό στην καθημερινότητά του. Άλλο ένα ενδιαφέρον και θα περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ελπίζω από τον Γενάρη φέτος θα έχουμε και ένα πολιτικό σύμβουλο στη δομή μας Αυτό το μείγμα πολιτικού λοιπόν και στρατιωτικού είναι νομίζω απόλυτα απαραίτητο για τη δομή μας. Επόμενη διαφάνεια. Ένα σχεδιάγραμμα, να θυμάστε ότι κάθε δύο χρόνια οι έξι στρατηγοί αλλάζουν. Αλλάζουν θέση και αυτός είναι άλλος ένας τρόπος να εκφράσουμε την βούλησή μας, να έχουμε ακριβώς πόλους εξουσίας που θα είναι σωστά κατανοημένοι μεταξύ των χωρών. Και χάρη διαφάνειας η Πολωνία θα αναλάβει την ηγεσία του Eurocorp το 2017. 19. Προπολογισμό 12-13 εκατομμύρια ευρώ. Περιορισμένο προπολογισμό 0,5% του προπολογισμού άμυνα του Βελγίου. 0,5%. Αρκεί βεβαίω για να δουλέψουμε σωστά υπό καλέ συνθήκε. Και ελπίζω ο προπολογισμό αυτό να παραμείνει σταθερό. Ένα ε, προπολογισμό χαμηλό και με την τιμή αυτή με την τιμή αυτή έχουμε ένα πλήρω σχεδόν εξοπλισμένο και, ε, και ε, εκπαιδευμένο επιτελείο και αυτό βεβαίω τονίζει και το γεγονό και υπογραμμίζει και το γεγονό ότι είμαστε και μια αποτελεσματική δομή. Και το υπογραμμίζω αυτό ω όρο. Αποτελεσματική δομή. Επόμενη διαφάνεια. Υλικό διαθέσιμο στο Eurocorp. Έχουμε container γραφεία. Έχουμε σκηνέ. Έχουμε ε, ε, γεννήτριες, έχουμε υπολογιστές, έχουμε πολλά. Και είμαστε το μοναδικό γενικό επιτελείο σώματος στρατού το οποίο συνδέεται με το ΝΑΤΟ και στην περίπτωσή μας βέβαια συνδέεται με την Ένωση που διαθέτει αυτό το υλικό μοναδική περίπτωση και αυτό το υλικό δεν ανήκει βεβαίω σε μένα αλλά στις χώρες πλαίσιο, δηλαδή σε εσά. Στους Γάλλους, στους Γερμανούς, στους Βέλγους, στους Λουξεμβούριου, στους Ισπανού, ε, Αυτό το υλικό ανήκει σε εσά η έδρα μας είναι στο Στρασβούργο, σε δύο κτίρια, το Πολύγωνο, όπως το λέμε. Το κοινοβούλιο είναι σε ωραία θέση, ωραία τοποθεσία στο κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς μας εξώθησαν εκεί, τέλος πάντων, στις κακόφημες περιοχές της ε, πόλης, αλλά τέλος πάντων, και εδώ δεξιά στη διαφάνεια βλέπετε το Λιζέ τοποθεσία δηλαδή που περιλαμβάνει το αρχή της υποστήριξης που έχουμε. Επόμενη διαφάνεια, ίσως πιο σημαντική διαφάνεια. Όταν έλαβα την ε, ηγεσία του Eurocorp, διαπίστωσα ότι η έννοια ε, χρήσης του Eurocorp ε, ήταν μιας δεκαετίας τουλάχιστον. Αναφέρθηκα σε ένα σώμα στρατού, το οποίο όμως ως έννοια μπορεί να μας κάνει να έχουμε λάθος εντυπώσεις. Δηλαδή, ε, δεν μιλάμε μόνο για επιχειρήσεις με 60.000 άντρες, εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο ως Γενικό Επιτελείο ε, πρέπει να είναι πολυχρηστικό, πρέπει να έχει δυνατότητα τέτοια πολυχρηστική και να είναι σε θέση να κάνει επιχειρήσεις σε κάθε ε, πιθανή κλίμακα φιλοδοξίας ή αξίας. Έχουμε βεβαίως στη, στην κορυφή πάνω ε, τις έντονες, τις σημαντικές επιχειρήσεις και κάτω έχουμε τις επιχειρήσεις, της δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευση κτλ. Δηλαδή έχουμε τις κούκλες, τις ρώσικες. Οι πιο μικροί είναι οι συνοδευτικές και υποστηρικτικές ε, επιχειρήσεις και οι πιο μεγάλοι βεβαίως οι κλασικές ε, επιχειρήσεις, οι συνήθεις με χιλιάδες, με συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτών. Έχουμε δύο κουτιά εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια το κουτί ή το τετράγωνο τέλο πάντων ΝΑΤΟ που καλύπτει, βλέπετε εδώ και τη σημαία, που καλύπτει τις πιο δύσκολες, τις πιο σκληρές αποστολές, ενώ εδώ η σημαία της Ένωσης καλύπτει τις πιο ευφυείς, όχι τις πιο επιές, γιατί ακούγεται άσχημα, αλλά τις πιο ευφυείς, τέλο πάντων, αποστολές, με προσέγγιση έτσι πιο παγκόσμια. Επόμενη, το μέλλον του Eurocorp. Όταν έλαβα εγώ το 2013, δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε μέχρι το 2020. Το 2020 και πάλι ε, θα βρισκόμαστε υπό το ΝΑΤΟ ως ε, μονάδα αντίδραση. Αλλά μέχρι το 2020 δεν είχαμε κανένα καθήκον. Εγώ λοιπόν έπεισα, ε, πιέζοντας, το υπεύθυνους άμυνα να κινητοποιηθούν ώστε να επανατοποθετήσουν το Eurocorp κάπου ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω τον κύριο Τανουσάν εδώ που με κοιτάει να επιθυμίσω ότι τότε προσπάθησα να πιστοποιήσω τους υπευθύνου άμυνα ότι αυτό πραγματικά ο σχέδιο ήταν ρεαλιστικό και θα έπρεπε να λάβει έτσι σάρκα. Έχουμε την αποστολή στο Μάλι. Το δεύτερο ΕΟΤ Μαλί, όπως λέγεται, στο δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτου έτους και θα έχουμε επίσης και ως Γενικό Επιτολείο ένα ρόλο το 2016 ο δεύτερο εξάμεινο ε, καλύπτοντας ένα σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ακολουθώντας και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Στο μέλλον το Eurocorp θέλουμε να θεωρείται ως το μοναδικό επιτελείο στρατού το οποίο θα είναι πολυχρηστικό και θα μπορεί να κάνει ε, επιχειρήσεις και ε, του ΝΑΤΟ αλλά και της Ένωσης. Επόμενη διαφάνεια. Δύο λόγια τελειώνοντας και κάποιες απόψεις σχετικά με το Eurocorp. Νομίζω ότι δεδομένη της νοοτροπίας, της κουλτούρας του Eurocorp και της πολιτικής του αξιοπιστίας από τα έθνη που το αποτελούν πέντε στην Πολωνία που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του πληθυσμού της Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματική απτή πολιτική βούληση. Αυτό που ελπίζουμε είναι στα πλαίσια των επιχειρήσεων που θα κάνει η Ένωση το Eurocorp να μπορέσει να μετατραπεί ε, στο γενικό επιτελείο του κανονικού στρατού, κανονικού στρατού που θα στέλνει στις αποστολές της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε αποστολές με, δια, διαφορετικό επίπεδο έτσι, στόχων και φιλοδοξίας και κάποιος είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να παρεμβαίνει παντού. Συμφωνώ απόλυτα με, αυτό, αυτή την άποψη. Το Africom που είναι μια αποκλειστικά και αμερικανική δομή στην Αφρική το Africom προσπάθησε να εγκατασταθεί στην Αφρική και πουθενά δεν τους αποδέχτηκαν και η έδρα του τώρα είναι στη Στουτγκάρδη. Το ΝΑΤΟ, κατά τη δική μου την απόψη και το όραμα, δεν είχε ποτέ την ε, ε, βούληση ή την δυνατότητα να παρενέβει στην Αφρική, που είναι εκτός τόπου, κατά την απόψη μου. Οπότε για τις μελλοντικέ απειλές, ε, Ανατολή, Ουκρανία, Ανατολική Ευρώπη κτλ. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά, εμείς οι Ευρωπαίοι, θα πρέπει βεβαίως να παρακολουθούμε ε, την Ανατολή μας σύμφωνα και σε συνεργασία με την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, αλλά θα πρέπει επίσης, επίσης να παρακολουθούμε στενά ε, αυτά που συμβαίνουν στη Βόρεια Αφρική, γιατί αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να εκτραπούν, ιδιαίτερα στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι η πρόκληση που έχει μπροστά της Ευρώπη στο μέλλον και το ΝΑΤΟ δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει στην Ευρώπη, στην Αφρική. Το Eurocorp συνοψίζοντας είναι ένα σώμα το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό και υποεκτιμάται. Βεβαίω έχει κατάλληλο υλικό, αλλά λείπει η πολιτική βούληση για την διάθεση στρατευμάτων στα πλαίσια μια διεθνού επιχείρηση. Χρειάζονται στρατεύματα, χρειάζεται στρατό και αυτή η δουλειά θα πρέπει να κάνει το Eurocorp. Ξέρω ότι, ξέρω ότι ίσως αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο σε κάποιες χώρες. Δηλαδή, αν υποχωρήσει το ΝΑΤΟ, θα μπορούσε μελλοντικά στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί το Eurocorp ως ένα έδος μόνιμου επιτελείου ευρωπαϊκού. Αυτό ε, σε κάποιους φαίνεται έτσι παράξενο και τους δυσαρεστεί Αλλά θα ήθελα να το πω αυτό. Τέλος, συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω, όπως λέμε στα αγγλικά, use it or lose it. Να το χρησιμοποιήσετε ή θα το χάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ähm, Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για τις ειλικρινείς παρατηρήσεις. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε με δεδομένη την πρώτο καθαδρία των πολιτικών επιλογών, αλλά πάντα είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τη δική σας αξιολόγηση, έστω και με διπλωματική διατύπωση. Πρώτος λοιπόν, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριος Μιχέλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Μπούξερ Σμιτ. για την παρουσίαση και τις θέσεις που διατυπώνεται, που ξέρω ότι δεν είναι απολύτως ε, συμπεφωνημένες προκαταβολικά με τα 28 μέλη του ΝΑΤΟ ή τα 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον των συναντήσεών μας. Χαίρομαι που μας εξηγείτε τι είδους δυναμικό μπορεί να έχει το Eurocore και που θα μπορούσε να αναλάβει δράση. Χάρη και στο μέγεθός του. Καθώς θεσμικά τουλάχιστον, με το επιτελείο του, είναι εδρεωμένο στο ΝΑΤΟ. Και άρα οιεσδήποτε συζητήσει και αμφισβητήσεις μπορούν να απαντηθούν πολύ γρήγορα εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Μπορεί λοιπόν το Eurocor να αναλάβει δράση για να εκπληρώσει κλασικές στρατιωτικές αποστολές ή εφόσον χρειάζεται να συνεργαστεί με τον ΝΑΤΟ. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή, όπως λέμε, να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Η εμπειρία προκύπτει και από τις πραγματικές αποστολές. Διερωτώ με λοιπόν εάν για τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου θα πρέπει να αναπτύξουμε και διεκδικήσεις σχετικές με το Eurocore. τι θα ήταν πιο καλό να είμαστε θέση να συστήσουμε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε σχέση με το Eurocore. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη μου ερώτηση. Κατά τα άλλα ελπίζω ότι με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη της πολιτικής βούλησης και φαντάζομαι και με την δραστηριοποίηση κάθε δυνατότητας που έχουμε στα χέρια μας και μέσω της νέας συνθήκης, αν και δεν είναι και τόσο πρόσφατη, αλλά εν πάση περιπτώσει η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει κάποιες δυνατότητες επιπλέον και μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για μια μόνιμη δομή, το Permanent Structured Cooperation, μια συνεργασία μόνιμα δομημένη που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια λειτουργούσα δομή που θα μπορούσε υπό συγκεκριμένε συνθήκε να αναλαμβάνει και δράση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την προοπτική, για τις συστάσεις, για τις ιδέες. Εμείς δεν καλούμε να λάβουμε αποφάσεις, αλλά ως κοινοβούλιο πρέπει και να δίνουμε ενάυσματα για σκέψη και να ελέγχουμε την εκτελεστική εξουσία. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Είναι διάλογος, αλλά όλοι πρέπει να καλυφθούν δύο μιλητές, δύο ερωτήσεις και ε, μπορείτε να απαντήσετε μετά. Ο Αντιπρόεδρος Τετίνα τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Κύριε Αντιστράτηγε, είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε σήμερα εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. Η παρουσίαση που κάνατε ήταν θαυμάσια. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα του Eurocall. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσφατα ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να αποσταλούν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε και στα στρατεύματα της ΕΕ. Μίλησε μάλιστα για αστυνομικές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Βεβαίως, εδώ είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ε, δεν σας θέτω συνεπώς το ερώτημα σαν πολιτικός, αλλά σαν στρατιωτικός. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν υπάρχουν στρατεύματα στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο τον ειρηνευτικό στην Ουκρανία. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Merci beaucoup, Monsieur le <laughs> Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ε, ερώτηση του κ. Γκέλλερ. Ε, όσον αφορά την ιστορία του Eurocore, βασικά είμαστε στραμμένοι προς το ΝΑΤΟ για κλασικές επιχειρήσεις. Βεβαίως, αν πάρετε ε, τα διάφορα είδη επιχειρήσεων από το Κωσυφοπαίδιο μέχρι το Αφγανιστάν, έχουμε περισσότερο σχέση με την ειρηνευτική δραστηριότητα με ένταση θα έλεγα. Όσον αφορά την διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου, αν μιλούσα προς τους πολιτικούς επικεφαλής μας, θα ρωτούσα, ξέρετε τι θέλετε, ε, μπορείτε να πετύχετε συνένεση ώστε να συνενώσετε τις αντιλήψεις σας για τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρώπης. Να είναι όλα αυτά περισσότερο συνεπή, να αντιληφθούν όλοι ότι η ασφάλεια του διπλανού είναι η ασφάλεια και του ίδιου. Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί κοιτούν προς τον Νότο και αντιμετωπίζουν όσο καλύτερα μπορούν την ροή των μεταναστών που αποβιβάζονται από τις αφρικανικές χώρες. Το φαινόμενο αυτό δεν ανησυχεί προς το παρόν τις βόρειες χώρες, αλλά μια μέρα οι μετανάστες αυτοί που θα έχουν αποβιβαστεί στις παραλίες του Νότου θα βρούνε τρόπο να περάσουν από ε, το Σέγγεν, να μπουν στο Σέγγεν και θα καταλήξουν στις βόρειες χώρες. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα μόνο για τη Λαμπεντούζα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόβλημα της Ουκρανίας και αυτό είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης. Βεβαίως η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες ανησυχούν περισσότερο άμεσα. Αλλά αν κοιτάξουμε τις οικονομικές συνέπειες, την παροχή ενέργειας, οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης μπορεί να πληρώσει τις συνέπειες μια μέρα. Ένας καλός τρόπος να πετύχουμε συνένεση πολιτική όσον αφορά τις απειλές και τα ζωτικά συμφέροντα είναι να θέσουμε όσον αφορά τις πληροφορίες και την στρατηγική ανάλυση το ερώτημα ποια είναι τα ζωτικά συμφέροντα του καθενός, της Ευρώπης και πώς μπορούν της Ευρώπης και του καθενός να συνδυαστούν ενδοεπισκόπηση λοιπόν στο επίπεδο το ευρωπαϊκό μια ανάλυση η οποία πρέπει να βασιστεί στη συλλογή βάσιμων πληροφοριών και την ανάλυση τους. Λοιπόν, όσον αφορά τους πολιτικούς ηθήνοντες, θα τους σύστηνα να δώσουν την προτεραιότητα στην πολυεθνικότητα και στην κοινή ομαδοποίηση των ε, μέσων, των εξοπλισμών. Παίρνω λοιπόν την Ισπανία, την Ιταλία κτλ. Ε, έχουν ένα αρχηγείο στο επίπεδο το στρατιωτικό ε, και δεν μπορούν να παράσχουν τα αντίστοιχα στρατεύματα. Μελλοντικά όμως θα είναι πολυεθνικές όλες οι επιχειρήσεις και πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη να δημιουργήσουν μια εθελοντική συμμαχία για την κοινή ομαδοποίηση, την οργάνωση των εξοπλισμών και των μέσων. Ε, υπάρχουν ειδικότητε βεβαίω και υπάρχουν καλά συστατικά σε κάθε χώρα ευρωπαϊκή. Στο Βέλγιο, παραδείγματο χάρη, μα αναγνωρίζουν διεθνώ ω ειδικοί για την εξουδετερώση ναρκών στη θάλασσα. Ε, υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν άλλες δυνατότητες. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι διαφορετικές δυνατότητες οργανωθούν κάτω από έναν επικεφαλής, τότε πετυχαίνουμε. Πολυεθνική διάσταση λοιπόν. Γιατί? Διότι όταν έχουμε σε ένα αρχηγείο ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς ορίζοντες, οδηγούμαστε έτσι σε εναλλακτικέ λύσεις όσον αφορά στο εθνικό δυναμικό, την στρατιωτική κουλτούρα και την ανάλυση της κατάστασης σε διάφορες χώρες. Η πολυεθνικότητα των αρχηγείων και των μονάδων μελλοντικά είναι το μέλλον της Ευρώπης. Τρίτο στοιχείο στην απάντησή μου και θα σταματήσω όσον αφορά μια μόνιμη δομή. Δεν είμαι τρελαμένος με αυτό, δεν θα είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνω. Κατά την άποψή μου Υπάρχουν πάρα πολλά αρχηγεία ε, σωμάτων στρατού. Και επειδή οι προϋπολογισμοί περιορίζονται σε το Eurocall σε 3, 5, 10 χρόνια, αν το ΝΑΤΟ αφαιρέσει τη συμβολή του στην άμυνα της Ευρώπης, σημαίνει αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε μόνιμα στην άμυνα και το Eurocore θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ενός μόνιμου αρχηγείου που θα είναι σε θέση να αναλύσει τα σχέδια, τις επιλογές κτλ. Και τώρα έρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Στετίνα. Η Ουκρανία είναι περίπλοκο θέμα. Για χρόνια ζήσαμε ε, ένα υπόδειγμα ειρηνευτικό, peacekeeping, peace force και άλλα διάφορα. Όλοι ήταν πεμπισμένοι ότι ποτέ ξανά δεν θα υπάρξει συμβατική ε, απειλή με τεθροκισμένα, πυροβολικό κτλ. Γι' αυτό ορισμένες χώρες έχουν τελείως εγκαταλείψει τα τεθεροκισμένα τους. Παραδείγματος χάρη το Βέλιο και έχουν εγκαταλείψει και την ιδέα να έχουν μέσα τα οποία επιτρέπουν εντατικές επιχειρήσεις. Κλειστήκαμε λοιπόν κάπως πρόωρα σε ένα σχήμα συγκρούσεων χαμηλής έντασης με βασικά τη διατήρηση της ειρήνης ή την αποκατάσταση της ειρήνης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι και πάλι αντιμετωπίζουμε μια χώρα που είναι έτοιμη για πολλά πράγματα. Το έχει αποδείξει ήδη. Κάνει, ε, είναι επικίνδυνο αυτό, σημαντικά επικίνδυνο για τον δυτικό κόσμο. Ο στρατιώτης που είμαι ε, σημαίνει ότι είμαι υπηρέτης ενός στρατιωτικού μηχανισμού που είναι στη διάθεση των πολιτικών. Ο πόλεμος είναι η κατάληξη της πολιτικής Συνεπώς, ε, η στρατιωτική δύναμη χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι στρατιωτικοί λοιπόν πληρώνονται για να παίξουν το ρόλο τους και να αναλάβουν τους κινδύνους. Ε, όλες οι δυνατότητες συγκρούσεων είναι ενδεχόμενες. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα λυθούν όμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε μία εισβολή των βαλτικών χωρών, παραδείγματο χάρη, με κινητικό τρόπο, αν μπορώ να το διατυπώσω έτσι. Ελπίδα μου είναι αυτό. Όσον αφορά τώρα τις αστυνομικές δυνάμεις δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Αλλά σε μια τέτοια κατάσταση πρώτα απ' όλα πρέπει να επιβληθεί η ειρήνη. Στη συνέχεια αρχίζει η ανοικοδόμηση του κράτους, των θεσμών, των φορέων, της εμπιστοσύνης στους φορείς, στους κρατικούς και στους πολιτικούς. Πρέπει να δημιουργηθούν και τα μέσα που επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν λογικά. Συνεπώς έχουμε μια φάση κρίσης. Μετά έχουμε μια φάση αποκατάστασης ειρήνης και στη συνέχεια ανασυγκρότησης. Όλα τα σενάρια παίζουν. Θα ήθελα το Ουκρανικό να λυθεί με τη διπλωματία και όχι σε μια εμπόλεμη ζώνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καν, ο κύριος Στογεύσκη, Νάρτ, Σεμπάλος. Και παρακαλώ να προβλέψετε αρκετό χρόνο ώστε να απαντήσει ο αντιστράτηγος. Μην κάνετε μακροσκελείς ερωτήσεις για να αφήσουμε χρόνο ώστε όταν χρειάζεται η διερμήνες να διακόψουν για το μεσημεριανό να έχει χρόνο να απαντήσει. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ τον στρατηγό για την εξαίρετη παρουσίαση και τα σχόλια. Με ενδιαφέρον ακούω τις ε, αξιολογήσεις σε σχέση με το soft power και το hard power. Ε, σε έναν κόσμο όμως που αλλάζει ταχύτατα η hard power, η σκληρή δηλαδή ε, άσκηση της ε, δύναμης που βρίσκεται, με περικοπές τους προϋπολογισμούς, που εντοπίζεται τη σχέση αυτή μεταξύ της σκληρής και της ήπιας δύναμης. Στο Ιευσκή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στρατηγέ μου. Έχω ορισμένε σύντομε ερωτήσει. Ποιε είναι οι προοπτικέ για τον προπολογισμό σα, ε, τον προπολογισμό του Eurocore δηλαδή, ω το 2020. Τι σχεδιάζετε, πώς μπορεί να βελτιωθεί η δημοσιονομική σας κατάσταση και δεύτερον σχεδιάζετε κάποια αποστολή στην Ουκρανία είτε ως εκπαιδευτική αποστολή είτε ως συμβουλευτική και τρίτον συμβάλλεται σε ένα βαθμό στην ε, ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη αναπτύσσει το Γαλιλαίος, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα και το Κοπέρνικους που είναι υπό ανάπτυξη. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό σε σχέση με τα ε, κινέζικα, τα ρωσικά, τα αμερικανικά συστήματα. Εγώ όμως νομίζω ότι θα πρέπει και οι, οι στρατιωτικές δυνάμεις να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός τέτοιου δορυφορικού συστήματος και θα ήθελα να παρακαλέσω και τη γραμματεία της Επιτροπής μας, τον κύριο Γκάλερ και λοιπούς συναδελφούς της Επιτροπής να προβλεφθεί η δυνατότητα να συζητηθεί και αυτό το θέμα σε μια συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Νάρτ. Ευχαριστώ, Στρατηγέ Μπούσενσμιτ. Ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε. Όμως έχετε πολύ το δίκιο. Είπατε ότι έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό στρατηγικής φύσης της ΑΧΕΛ που πέρα από στρατιωτική σύραξη είναι ένα θέμα κοινωνικό. Για τους γνώστες της Σαχάρας εδώ και 10 χρόνια ξέρουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα εμφανιζόταν κάποια στιγμή αλλά αυτό που βλέπω εγώ και ελπίζω να μου απαντήσετε είναι ότι εμείς δίνουμε μια ακατάλληλη απάντηση. Η μοναδική απάντηση που δίνουμε στο, στη Σαχέλ είναι μέσω Γαλλίας με τις επιχειρήσεις Ερβάλ και Παρκάν και έστω ε, και δεν αφορά άμεσα την ε, Σαχέλ έχουμε την Μπόκο Χαράμ, το στρατό του Τσάτ και το στρατό της Γαλλίας. Εγώ ήμουνα στο Μάλι τα Χριστούγεννα παρατηρητής στην αποστολή της, την εκπαιδευτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι τελείως τυχαία. Μετά από ένα έτος εκπαίδευσης στο Μάλι δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ούτε καν ένα λειτουργικό λόγο. Για να μην σας πω για ταξιαρχίες κλπ. κλπ. Και η απόδειξη είναι ότι όταν συγκρούονται τα στρατεύματα του Μάλι είναι τελείως άχρηστα και τους νικούν κατά κράτος οι αντίπαλοι. Η εκπαίδευση είναι ανεπαρκής, με ανεπαρκές υλικό και σε κάποιες περιπτώσεις είναι χωρίς υλικό γιατί δεν έχουν στη διάθεσή τους όπλα. Εγώ έμενα με το στόμα ανοιχτό όταν είδα ότι το γερμανικό στράτευμα εκπαίδευε το στρατό του Μάλι στην έρημο και τους εκπαίδευαν στην διάβαση ποταμών. Ποτάμια δεν υπάρχουν στην έρημο. Και ό,τι υπάρχει το έλεγχε ο γαλλικός στρατός. Οπότε πώς γίνεται μπροστά σε αυτό το μεγάλο στρατηγικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη εμείς να δίνουμε απαντήσεις τόσο ακατάλληλες μετά αφού μετά από ένα έτος δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ούτε καν έναν λειτουργικό λόγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα υπόλοιπα είναι η ουτοπία. Έχουμε ακόμα την κυρία Σεμπάλο, την κυρία Γκόμες. Παρακαλώ, η κυρία Σεμπάλο πρώτα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά. πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα ποια είναι η σχέση με τη Λαμπεντούζα και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Εγώ είμαι Σουηδή. Και η Σουηδία είναι από τις χώρες που δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημά σα. Ίσως κάτι να κατάλαβα λάθος όμως. Και επίσης, άκουσα τα τελευταία λόγια του στρατηγού. Use it or lose it. Χρησιμοποιήστε το ή αλλιώς θα το χάσετε. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο το Eurocore σε επιχειρήσεις για την ειρήνη Φερρυπίν των Ηνωμένων Εθνών, για υποστήριξη κρατών της Αφρικής. Υπάρχει τέτοια ανάγκη. Και μπορείτε εσείς να το αναλάβετε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Η ερώτησή μου, μετά τα όσα είπε ο κύριος ε, Καν για την ε, ήπια και τη σκληρή δύναμη. Θεωρείτε ότι η κατάσταση στρατηγικά σε σχέση με το συμβαίνουν στην ε, Ουκρανία έχει αλλάξει ως προς τη ε, μελήματα για τη χρήση της πυρηνικής ε, απειλής. Γιατί ξέρετε ότι έχει υποβαθμιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια και κάποιοι θεωρούν ότι είναι αντιπαραγωγική η επισήμανση της, του πυρηνικού οπλοστασίου. Το peacekeeping mode στο οποίο αναφερθήκατε, λειτουργία διατήρησης της ειρήνης. Μια και ακριβώς αυτό ζητάει το PKO όπως το λέμε, η Ουκρανία. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να μην χάσουμε όπως λέγατε το δυναμικό που έχουμε. ο Πρόεδρος. Στρατηγία, όπως βλέπετε, με τους ε, πολιτικούς μπορείτε, αν δεν είστε υποχρεωμένος όμως, να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ναι, θα απαντήσω, αλλά όχι με τη σειρά που ακούστηκαν, αλλά με μια σειρά αύξουσα δυσκολίας των ερωτήσεων. Και θα απαντήσω πρώτα στον Πολωνό βουλευτή. Είναι ευνοϊκές οι προβλέψεις και αισιόδοξε για την χρηματοδότησή μας. Προς το παρόν αρκεί ο προϋπολογισμός μας, πρώτον, και δεύτερον δεν έχω κανένα σημείο ή μήνυμα ότι μπορεί να μειωθεί. Βεβαίως θα χρειαστεί η Πολωνία να αναλάβει σημαντικό ε, σημαντική επιβάρυνση με την έννοια ότι εντάσσεται στο Eurocore με 100 άτομα προσωπικού αφενός, αφετέρου δε, καθώς ενισχύει την παρουσία της και στο σώμα, το βορειοανατολικό σώμα του Στετίνα. Άρα όλα αυτά θα κοστίσουν χρήμα στον Πολωνό φορολογούμενο. Αλλά για μας προ, προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει ένδειξη περί περικοπών στον προϋπολογισμό. Για αποστολές εκπαιδευτικέ στην Ουκρανία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη προς το παρόν. Όλα αυτά πιστεύω ε, θα έπρεπε να ενταχθούν σε μια διαδικασία που θα ήταν ούτως ή άλλως πολύ περίπλοκη. Θα έπρεπε να προσδιοριστούν ε, οι διαδικασίες ετυπώσεις εργασία ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη. Περίπλοκα όλα αυτά και... Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από εμά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, δεν έχουμε προλάβει τις εξελίξεις. Για ένα δορυφορικό σύστημα ομολογώ άγνοια και αναρμοδιότητα δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα το οποίο μας καλύπτει, υφίσταται δηλαδή αυτή η δορυφορική, αυτό το δορυφορικό δυναμικό, ε, δεν υπάρχει πρόθεση να ενισχυθεί. Η... Για την ερώτηση του κ. Νάρτ, Θα αναφερθώ και πάλι στην εμπειρία μου από την ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για να αναφερθώ στο, στην επιχείρηση εκπαίδευση στο Μάλι. Δεν ξέρω γιατί πάντα θεωρείτε ότι για να, για να σταθεί στα πόδια του ένα χαμένο κράτος, ένα αποτυχημένο κράτος, failed state, μπορεί να χρειαστούν έξι μήνες. Όχι. 20 χρόνια ίσως και περισσότερο. Μια με δύο γενιές χρειάζεται. Μια αποστολή λοιπόν η οποία έχει διαρκέσει έξι μήνες, ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, δεν περιμένουμε ότι θα έχει σαφή, ξεκάθαρα, ορατά αποτελέσματα. Για το Μαλί ούτως ή άλλως, μια και θα πάει στο δεύτερο εξάμεινο του 2015 το Eurocore, θα έχω την ευκαιρία εγώ να επανέλθω και να το ξαναδώ. Ο Γερμανός στρατηγός ε, που ηγείται της αποστολής, επιφορτισμένος με την αποστολή όπως λέγεται, ένας άνθρωπος με πολύ πρακτική θεώρηση των πραγμάτων, είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει να εξασφαλίσει τα μέσα που θα αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μέσα μηχανικά για την για να μπορούν να διασχίζουν οι Μαλιανοί ε, μεγάλα ποτάμια, ίσως να μην είναι η πρώτη προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει, ε, οι παράγοντε επιτυχία θα είναι οι εξή για την αποστολή. Να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και πλαισίωση, την συντήρηση με τον χρόνο, να διατηρηθεί δηλαδή σε υλικό αλλά και σε εντολή. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να εκπαιδεύουμε στρατιωτικούς οπουδήποτε στον κόσμο να τους φτάνουμε σε ένα επίπεδο ικανότητας και μετά να τους τραβάμε την ε, ανεμόσκαλα κάτω από τα πόδια και να λέμε τι κάνουμε, φεύγουμε. Όχι, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό πιο μακροπρόθεσμο, 5, 10, 15, 20 χρόνια ακόμα. Δεύτερη επιτυχία για να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, ε, την επιτυχία αυτής της αποστολής κατάρτισης, εκπαίδευσης, πρέπει να αμείβονται οι στρατιωτικοί. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο στο πρώην Βελγικό Κονγκό, τη λάψους ήταν αυτό που διέπραξα, ε, την ε, πληρωμή την είχε αναλάβει η διοίκηση του στρατού. Δηλαδή η Κινσάσα έστελνε στον περιφερειακό διοικητή το χρήμα και αυτό το μοίραζε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό βέβαια, το σύνδρομο του της πυραμίδας ε, των ποτηριών σαμπάνιας στις δεξιώσεις. Δηλαδή το πρώτο ποτήρι παίρνει πολύ υγρό ενώ τα τελευταία μένουν άδεια. Αυτό συνέβαινε και στη διαχείριση της αλυσίδας πληρωμών ε, στην Κινσάστα. Πρέπει η διαχείριση αλυσίδας πληρωμών να είναι διαφορετική από την αλυσίδα διοίκησης και στο Μαλί όπως παντού όπως δεν συμβαίνει σε όλα τα αφρικανικά κράτη. Ξέρουμε ότι στη ζωή του στρατιώτη έχει πρωταρχικό ρόλο η οικογένειά του. Εάν δεν λαμβάνουμε υπόψη την οικογένεια του στρατιώτη, ο στρατιώτης δεν θα είναι ποτέ καλός στρατιώτης. Με όλους αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα, μπορούμε σε ένα αφρικανικό κράτος να εξασφαλίσουμε έναν στρατιώτη γερό, δυνατό, ε, θαραλέο, πατριώτη. Όλα αυτά όμως το επαναλαμβάνω χρειάζονται χρόνο και μέσα. για την κυρία Σέβαλο. Λαμπεντούζα. Κοιτάξτε, ο καθένα έχει τη δική του θεώρηση των πραγμάτων. Οι δικέ μου προβλέψεις και ελπίζω να αποδειχθώ ψεύτης είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές που ξεκινούν από ορισμένα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο θα γίνουν πολύ σύντομα ανεξέλεγκτες. Και όπως είπα ελπίζω να βγω ψεύτης θα δούμε χιλιάδες μεταναστών να ξεμπαρκάρουν στις ακτές μας. Στο καλέ τώρα περιμένουν 3.000 για να περάσουν στο Νήμανο Βασίλειο. Ο χώρος του Σέγγεν είναι ανοιχτός χώρος. Όποιος θέλει ταξιδεύει όπου θέλει ή σχεδόν. Ε, οι μεταναστευτικές αυτές ροές θα αγγίξουν περισσότερο ή λιγότερο τα ευρωπαϊκά κράτη. Και δεν πρέπει να ε, βλέπουμε με όρους ε, απόλυτους στο μετανάστη ως κάποιον ε, που μπορεί να είναι επιζήμια παρουσία. Κάποιοι ναι, αλλά κάποιοι άλλοι έρχονται μαζί με την ελπίδα τους και τη δυστυχία τους και μπορούν να αποτελέσουν μια θετική συμβολή. Άρα χρειάζεται μια μεταναστευτική πολιτική πραγματικά ευρωπαϊκή και όχι εθνική. Κύριο παράδειγμα αποτυχίας ε, πολιτικής είναι η διαχείριση των μεταναστών στο καλέ μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Είναι απαράδεκτη και αποτρόπαιη εικόνα. Αυτά όσον αφορά τη Λαμπεντούζα. Για το Eurocore, αξιοποιήστε το ή θα το χάσετε. Use it or lose it. Δεν νομίζω ότι είναι ένα μέσον που μπορούν να αξιοποιήσουν τα Ηνωμένα Έθνη το Eurocore. Είναι μια λύση πολλαπλή. Μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές δομές αλλά όχι μόνο για, δομές, για αποστολές ε, μικρής ή πολύ μικρής έντασης, αλλά και για αποστολές, υψηλής, υψηλές, υψηλής έντασης, όπως ε, η αποστολή Άρτεμι το 2003. Τη στιγμή που έχουμε μια πολιτική επιλογή, βούληση, και τη στηρίζουμε με τα κατάλληλα στρατιωτικά μέσα, στρατιωτικό προσωπικό, μπορούμε να προλάβουμε μια κατάσταση και να τη σταθεροποιήσουμε πριν εκραγεί. Το πρόβλημα είναι με την Αφρική, με την ε, περιοχή του Σαχέλ, με τη Λιβύα, με το Μαλί, είναι ότι καθυστερούμε πολύ στην ανταπόκριση. Πρέπει να κοιτάξουμε την αιτία και όχι τη συνέπεια. Συνέπεια είναι Λαμπεντούζα. Αιτία όμως είναι το Σαχέλ, είναι η αταξία, είναι οι ακρότητες, είναι οι ε, φανατισμοί και οι ριζοσπαστισμοί. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο πρέπει στη βάση του να καταπολεμήσουμε με μέσα στεναρά και θα επανέλθω εδώ στην απάντηση που έδωσα στον ε, βουλευτή νωρίτερα για το hard και το soft power ότι ώρες, ώρες δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αξιοποιήσουμε τη σκληρή δύναμη hard power του φέκια και κανόνια. Με λύπη μου το λέω, αλλά αυτό που έκανε η Γαλλία για να αποκαταστήσει κάποιο είδου τάξη σε ορισμένες αφρικανικές χώρε ήταν, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε, πίσω από το δάχτυλό μα, ήταν στρατιωτικέ επιχειρήσει, πολεμικέ επιχειρήσει. Και αυτό το λέω γιατί σε ορισμένε περιπτώσει είναι η κατάσταση τέτοια που δεν υπάρχει διαπραγματευτή. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γιατί δεν υπάρχει διαπραγματευτή. Δεν υπάρχει κανεί με τον οποίο να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με την ΤΑΕΣ γιατί δεν υπάρχει ε, συνομιλητή καταλαβαίνουν μόνο ένα πράγμα, το τουφέκι στο κεφάλι. Άρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Άρα, στην ερώτηση hard και soft power, πολύ καλά, εφόσον βέβαια δεν είναι υπερβολική η αντίδραση. Πολλές φορές όμως οι συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια αποδεικνύεται ότι δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της διπλωματίας ως μέσον, γιατί δεν μπορεί κανείς να συνδιαλλαγεί, αλλά είναι αναγκαία η βίαιη παρέμβαση με στρατιωτικά μέσα στις στις περιοχές που βεβαίως ασφαλώς θα φέρουν και ζημιές. Άλλη μια ερώτηση την οποία δεν έχω απαντήσει για την κυρία Γκόμες και την Ουκρανία. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω, δεν έχω αρμοδιότητα να απαντήσω για το πυρηνικό. Είναι περίπλοκο ζήτημα, δεν τολμώ ούτε να τα αγγίξω. Αυτό που έχει αλλάξει όμως ως προς την αντίληψη των ε, δυτικών κρατών σε σχέση με την Ουκρανία και ακροθυγώς το ανέφερα νωρίτερα, είναι ότι δεν βρισκόμαστε πλέον σε mode ότι όλα καλά, όλα ωραία. Δεν είμαστε δηλαδή σε διάθεση ε, να ρυθμίζουμε τα ζητήματα πάντοτε με ε, την ε, διατήρηση της ειρήνης και τον εφησυχασμό. Μερικές φορές αυτό δεν φέρνει αποτελέσματα. Το ζήτημα λοιπόν της Ουκρανίας σε σχέση με τα δυτικά κράτη έχει την εξή σημασία ότι καθιστά σαφέ στους αρμόδιους για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων ότι αν αφήσουν να καταστραφεί ένα εργαλείο που έχουμε στη θέση μας αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή καταστροφή, θα βρεθούμε κάποια στιγμή ε, να το χρειαζόμαστε και τότε η μόνη λύση που θα έχουμε στη θέση μας θα είναι να στραφούμε στο ΝΑΤΟ. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή να έχει στα χέρια της επαρκή στρατηγική αυτονομία ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την αναγκαία της ασφάλεια. Αυτό είναι το tipping point, το σημείο ρήξος δηλαδή των θέσεων και των επιλογών που μπορούν να έχουν οι δυτικέ χώρε σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει ή τι πρέπει να γίνει στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας. Θα ήθελα να υποφεληθώ της ευκαιρία που έχω το λόγο για να ευχαριστήσω και πάλι τον στρατηγό μας. Τον ευχαριστώ που μας παρουσίασε μια πολύ ρεαλιστική αντίληψη ενός στρατιωτικού. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τους πολιτικούς να μπορέσουν να έχουν και μια διαφορετική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασής μας, επόμενη συνεδρίαση 16 Μαρτίου εδώ στις Βρυξέλλες. Γεια σας.